La séance est ouverte. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ε, ενημερώσω για ορισμένα νέα. Καταρχάς για την απόφαση των συντονιστών της 24 η Σεπτεμβρίου. Βρίσκεται στο φάκελο με τα έγγραφα της συνεδρίασης και αν δεν έχετε αντιρρήσεις θεωρώ ότι εγκρίνονται οι αποφάσεις των συντονιστών. Να σας επιθυμίσω τα εξής για την ημερήσια διάταξη και τον προϋπολογισμό τις επόμενες εβδομάδες. Την 5η 18 Οκτωβρίου από τις 10 ως τις 11 ώρα το πρωί τα μέλη είναι προσκεκλημένα να συμμετάσχουν σε μια διοργανική συνεδρίαση για τις πληρωμές παρουσία Επιτρόπου Έτιγκερ παρουσία εκπροσώπου της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος και ποιοι θα απαρτήσουν τις υπόλοιπες αντιπροσωπείς του Συμβουλίου. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια έκθεση για τις προβλέψεις, για τις πληρωμές και τα έσοδα από σήμερα μέχρι και το 2023. Ένα έγγραφο εξαιρετικά σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη ε, το εύρος των υπολείπων προς εκαθάριση, που είναι περίπου 280 δις δηλαδή πάνω από μια μισή φορά ο δικός μας προϋπολογισμός. Ξέρετε ότι στις 18 Οκτωβρίου θα γίνει τριμερής διάλογος για θέματα προϋπολογισμού σε, στην Επιτροπή και κλεισμένων των θεϊρών για να υπερασπιστούμε τις τροπολογίες που εγκρίναμε στην Επιτροπή για τον προϋπολογισμό πριν από δύο εβδομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα Έχουμε τη δική μας πρόταση για τον προπολογισμό του 2019 και θα συζητηθεί την επόμενη συνεδρίαση της ομάδας μας στις 24 Οκτωβρίου. Θα ψηφίσουμε και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η περίοδος συνδιαλλαγής. Ορισμένα μέλη της Επιτροπής μας θα οριστούν από τη δική τους πολιτική ομάδα για να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Άρα αυτά τα μέλη καλούνται να σημειώσουν ότι η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής θα λάβει χώρα την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί. Η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, όπου μάλλον θα κλείσουν οι διαπραγματεύσεις, εκεί δίνανται να ε, κλείσουν οι διαπραγματεύσεις, θα γίνει την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Και σημειώνουμε ότι Παρασκευή 16 Νοεμβρίου είναι μετά από την εβδομάδα της Ολομέλειας του Στρασβούργου. Ελπίζω να μπορούμε να κλείσουμε την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, εάν όμως στις 8 το βράδυ δεν έχουμε την πεποίθηση ότι κλείνουμε με ικανοποιητικό τρόπο, τότε θα κηρύξω τότε τη λήξη της συνεδρίασης και θα τα ξαναπούμε στις 19 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Ιδού λοιπόν τα νέα και τη, τα μελούμενα τα οποία ήθελα να μάθετε και να γνωρίσετε. Έχετε λάβει μία ανακοίνωση για τα πρακτικά της συνεδρίασης που έλαβε χώρα στις 29 Αυγούστου και λογικά τα έχετε διαβάσει αυτά τα πρακτικά. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά της συνεδρίασης της 29 Αυγούστου. Η δική μας συνεδρίαση τώρα λαμβάνει χώρα σε ένα ιδιαίτερο υπόβαθρο, διότι ο συνάδελφος Τόρβαλτς συνοδεύεται από έναν αναπληρωτή βουλευτή και μπορεί να μας τον παρουσιάσει το μέλος. Να μας την παρουσιάζει. Σας ευχαριστώ. Με λένε Άνεκβεν Χβάρα, είμαι 16 ετών, είμαι από τη Φιλανδία και έρχομαι σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι λαμβάνω μέρος σε μία δράση για την ημέρα κατά την οποία τα κορίτσια αναλαμβάνουν και ασκούν τα δικαιώματά τους σε συνεργασία με ομάδες για τα δικαιώματα των παιδιών. Είναι η Διεθνής ημέρα των κοριτσιών. Έχουμε Girls Takeover, αυτό το και έτσι μπαίνουμε στη θέση ηγετών πολιτικών που λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις. Ε, καθόμαστε στην καρέκλα τους αν θέλετε και παίρνουμε τη σκητάλη ως ε, μια δράση ενδυνάμωσης. Και είναι το κάλεσμα και η έκκληση που απευθύνουμε για έναν κόσμο με περισσότερη ισότητα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία σας ακούσαμε Αναπέλ και σας χειροκροτούμε. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας υποδέχεστε εδώ, λέει ο κύριος Τόρβαλτς. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανέλαβαν τα ενία και τη σκητάλη τα κορίτσια. La relève est assurée. Maintenant, je donne... Πράγματι, η συνέχεια στο έργο μας έχει εξασφαλιστεί. Να δώσω το λόγο για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Η κυρία Καρτία Θαμπάλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσουμε με τις ε, καθημερινές εργασίες, ε, να σας πω ότι η υπηρεσία επικοινωνιών δουλεύει πολύ καλά και μας είπε ότι την Κυριακή ήταν τα γενέθλιά σας και το μάθαμε και θέλουμε να σας ευχηθούμε ολόψυχα ε, χρόνια πολλά να τα χιλιάσετε. Voilà qui me touche au plus, plus... Ο Πρόεδρος, με συγκινείτε, με συγκινείτε βαθύτατα. Δυστυχώς δεν με κάνετε πιο νέο από ότι είμαι, αλλά μου δείτε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και δέχομαι ε, την παρέμβασή σας ως ένδειξη βαθιάς φιλίας. Ε, τρέφω μεγάλη εκτίμηση και ε, θερμές ευχαριστίες προς το πρόσωπό σας. Είναι παρακαλώ. Και εγώ θέλω κύριε Πρόεδρε να σας ευχηθώ. Ελπίζω να μείνετε όπως είστε για να είστε πάντα ευτυχείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, έκθεσή μου για την κινητοποίηση του Ταμείου της Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή βοήθεια στη Λετωνία είναι μια έκθεση που ουσιαστικά αφορά την αλληλεγγύη, που είναι και ένας από τους ακρογωνίους λίθους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τις αρκετές δυσκολίες και κρίσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να παρέχει βοήθεια στα κράτη-μέλη της εφόσον υπάρχει κάποια κατάσταση ανωτέρας βίας. Ίσως γνωρίζετε πως πέρυσι από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο η Λετωνία βίωσε άνευ προηγουμένου βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Με αποτέλεσμα ολόκληρη χώρα να πληγεί σοβαρά, αλλά πρώτα απ' όλα μια από τις πιο όμορφες αλλά και λιγότερο ευνεμένες ε, ανατολικές περιφέρειες Λότκαλ λέγεται με πάρα πολλές ζημιές πάνω από 380 εκατομμύρια ευρώ ε, για μια μικρή χώρα σαν τη δική μας ε, με 2 εκατομμύρια κατοίκους μόλις. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ οδυνηρό. Οι συνολικές ζημίες ε, είναι διπλάσιες ε, του ε, ορίου των 145,7 εκατομμυρίων ευρώ που είναι το κατόφλι για να αναγνωριστεί μια καταστροφή ως μείζον φυσική καταστροφή διπλάσια στις ζημίες. Λοιπόν, επομένως επιλεξιμότητα υπάρχει για την παροχή βοήθειας διαμέσου του Ταμείου Θέλω να σας αναφέρω τον αντίκτυπο των πλημμυρών το 2017 ε, το μεγαλύτερο μερίδιο του κόστου αφορούσε το σύστημα αποχέτευσης ε, και αποστράξη και τι σχετικέ υποδομέ στο δημόσιο. Υπήρχε όμως και πολλή ε, ζημιά για τη γεωργία. Χάσαμε καλλιέργειες και η γεωργική, το γεωργικό σύστημα αποχέτευσης είχε με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο σύστημα προστράγγισης, στι δρογικές εγκαταστάσει, στα φράγματα, στι μεταφορές και σε πολλέ άλλες υποδομές. Και στο σιδηροδρομικό δίκτυο 184 αυτοκινητόδρομοι υπόστησαν ζημιές και οι συνδρομικές συγκοινωνίες διακόπηκαν προσωρινά. Ε, κηρύχθηκε η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ε, υπήρχαν προβλήματα στο να λειτουργήσουν σωστά και οι κρατικές υπηρεσίες, πλημμύρισαν και σχολεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες έπρεπε να κλείσουν και από προσωπική εμπειρία. Εγώ κολύμπαγα εκεί που πριν ήταν χωράφια. Με την οικογένειά μου πήραμε το, ε, τη βάρκα και πηγαίναμε πάνω πλέαμε σε ένα χωράφι σίκαλης, προηγουμένως δηλαδή. Και ε, πάνω, από 17,7 εκατομμύρια κατά την κρίση της Κομισιόν θα πρέπει να κινητοποιηθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης προς ε, τη Λετωνία. Και θέλω να τονίσω ότι δεν θα χρειαστεί τροποποιητική διορθωτική επιστολή για τον ε, προϋπολογισμό. Γιατί θα καλυφθεί από το φετινό ε, προϋπολογισμό η συμβολή από το ταμείο είναι μόνο το 5% ε, των ε, ζημιών. Παρ' όλα αυτά, από το 2002 που εισήχθη αυτό το ταμείο και δίνει βοήθεια στα κράτη-μέλη που βρίσκονται πολύ σε αστραϊκή κατάσταση, γιατί δεν γνωρίζει ε, σύνορα τεχνητά η φύση, αυτή είναι η πιο προφανής, η πιο ορατή βοήθεια και καταδεικνύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας τους Ευρωβουλευτές αυτές είναι οι περιστάσεις που μας βοηθούν να δείξουμε ότι πραγματικά βοηθάμε τους ενδύεις. Γι' αυτό ζητώ την κινητοποίηση αυτού που Ευχαριστώ. Είναι κοινό ευρωπαϊκό αγαθό ελεγγύη, λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε κυρία Συγγήτρια. Περνάμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Καρίν Γκλοενέκ Μογά. Ήρθατε μόλις, έχετε, θέλετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα συμφωνήσω με τα λέγατε της ηγήτριας. πως είναι προφανές, θεωρώ και εγώ ότι η αλληλεγγύη είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρακολουθήσω με προσοχή τα έργα και θα παρακολουθούμε την κατάσταση και η ομάδα μου και εγώ προσωπικά. Πρόεδρος, δεν βλέπω να είναι παρόν κάποιος άλλος και έτσι Επιθυμεί κάποιος άλλος συνάδελφος να λάβει το λόγο. Αν όχι, ολοκληρώνουμε εδώ. Η συγγήτρια ήταν τόσο πιστική που δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε άλλο. Θα ήθελα να σας αναφέρω ε, ότι υπάρχει με κατάθεση τροπολογιών... Α, όχι. Ναι. Ναι. 11 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 5 Νοεμβρίου και η Ολομέλεια του Νοεμβρίου στο Στρασβούργο, η πρώτη Ολομέλεια του Νοεμβρίου στο Στρασβούργο, είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί σε εκθέσεως αυτής. Και τώρα θα περάσουμε στην ενδιάμεση έκθεση για το πι δελτα πι. Μίζων έκθεση ε, όπου παίρνει θέση το Κοινοβούλιο εν της προσεχούς συμφωνίας και για το πι δελτα πι για τους ιδίους πόρους. Μια μισή ώρα περίπου προβλέπεται ε, για τη συζήτηση του θέματος αυτού. Θα ακούσουμε και του συζητητέ από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Του ευχαριστώ που είναι εδώ παρόντες και δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στους δικούς μας συνεισηγητέ. αλλά ψάχνω να την Ιζαμπέλ Τόμα. Α, εκεί είναι, μάλιστα. Στου συνεισηγητέ, λοιπόν. Δεν ξέρω, Γιάννη Όλμπριχτ θα πάρει πρώτα το λόγο ή η Ιζαμπέλ Τόμα. Η Ιζαμπέλ Τόμα, λοιπόν. Ναι, θα εναλλαχθούμε με τον ε, Γιάννη Όλμπριχτ. Θα δούμε πώς θα πάει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, η Επιτροπή μας αποφάσισε να να ετοιμάσει, να συντάξει την ενδιάμεση έκθεση για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο βάσει της τακτικής διαδικασίας μετά το ψήφισμα του περασμένου Μαΐου, δηλαδή Ιουνίου. Αποφασίσαμε να το πράξουμε αυτό βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως προβλέπει η τακτική διαδικασία αλλά και βάσει της εντολής, της διαγματευτικής εντολής που μας ανατέθηκε τον Μάρτιο του 2018. Διότι στην έκθεση πρωτοβουλίας τον Μάρτιο του 2018 διευκρινιζόταν ότι πρόκειται για διαπραγματευτική εντολή για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επιμένω στο γεγονός ότι τον εργαστούμε στη βάση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της έκθεσης του Μαρτίου μας οδήγησε στις εξής δύο αποφάσεις. Πρώτη καινοτομία. Βασιστήκαμε στην έκθεση σαν ήταν έκθεση συναπόφασης για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο. Άρα τροποποιήσαμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή υποβάλαμε τροπολογίες αν για μια οποιαδήποτε έκθεση και δεύτερη αλλαγή που αποφασίσαμε να επιφέρουμε είναι οι αριθμοί, τα αριθμητικά στοιχεία, με ένα πίνακα με όλα τα αριθμητικά στοιχεία για όλα τα προγράμματα. Αυτό χάρη στην πείρα της διαποτευτικής ομάδας αυτών που διαπραγματεύτηκαν το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο και επειδή μα είπαν ότι οι διαπραγματεύσει ε, για τα αριθμητικά στοιχεία συνήθω είναι οι πιο δυσχερεί. Η έκθεση αυτή λοιπόν συμπερι... Ε, συμπεριλάμβανε δύο καινούργια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα την ε, έκθεση που ήταν σαν έκθεση συναπόφαση και μετά το σύνολο των αριθμητικών στοιχείων για όλα τα προγράμματα. Ω προ τη μέθοδο που ακολουθήσαμε πέραν των δύο αυτών καινούργιων στοιχείων, όπω θα ξέρετε, δεν είναι δικό μα ρόλος, δική μας αρμοδιότητα, να αποφασίσουμε εκ μέρου των άλλων συνυπεύθυνων επιτροπών, όμως στην έκθεση του Μαρτίου υπήρχαν δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, κόκκινες γραμμές απαγορευτικά όρια που ήταν εύκολο να μεταφραστούν σε τροπολογίες επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέσα στον πίνακα. Για παράδειγμα, ότι ψηφίσαμε ότι πρέπει να τεπλασιαστεί η πρικοδότηση του Εράσμους ή ότι πρέπει να διπλασιαστεί αυτή του κόσμου ή την, ε, για την Youth Initiative πάλι, διπλάσιο ποσό ή ότι πρέπει να προφυλάξουμε την ε, συνοχή, τη γεωργία. Εκεί δεν υπήρχε δυνατότητα διαφορετικής ερμηνείας. Πήραμε την έκθεση, υποβάλαμε τις σχετικές τροπολογίες και τα αριθμητικά στοιχεία τα συμπεριλάβαμε στον πίνακα, όπως προέκυπταν. Αυτό ήταν το απλούστερο. Όμως στην έκθεση του Μαρτίου υπήρχαν και άλλα στοιχεία. Λόγω χάρη ένα νέο πρόγραμμα όπως η εγγύηση για τα παιδιά, το Child Guarantee ή όταν έλεγε ότι ένα πρόγραμμα at least τουλάχιστον θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο που προβλεπόταν αρχικά. Δηλαδή, ας πάρει περισσότερα, αλλά μην το αποκλείσουμε κιόλα. Κοιτάξαμε τα ακριβή ποσά που ίσχυαν και είδαμε αν μπορεί να υπάρχει κάποια αυξητική πρόοδος. Για ό,τι ήταν σαφές ξεκάθαρο και ξάστερο στην έκθεση του Μαρτίου, λοιπόν, απλώς τα μετατρέψαμε σε αριθμητικά στοιχεία και σε τροπολογίες. Ό,τι μπορούσε να ερμηνευτεί διαφορετικά, το παραπέμψαμε στις αρμόδιες επιτροπές. Έτσι, καλέσαμε τις συνυπεύθυνε επιτροπές να εργαστούν βάσει της έκθεση για γνωμοδότηση του Μαρτίου 2018. Με τον Γιάν οργανώσαμε δύο-τρεις, δεν τώρα, συνεδριάσεις με του υπεύθυνου συζητητέ από τις ε, συνυπεύθυνε επιτροπές και του ζητήσαμε τις συνεισφορές τους, αριθμητικά στοιχεία έστω, πριν συντάξουμε την έκθεση. Κάποιοι πρόλαβαν Άλλοι καθυστέρησαν. Άλλοι δεν ξέρω αν θα μα στείλουν κάποτε κάτι, είναι ένα μυστήριο για μένα. Αλλά πιστέψτε με, εμεί κάναμε ό,τι παίρνει από το χέρι μα. Και εδώ και στι πολιτικές ομάδε και στι ε, επιμέρους επιτροπέ για να μα στείλουν τι απόψει του. Υπάρχουν κάποιε προσαρμογέ που πρέπει να γίνουν βέβαια. Βάσει των όσων θα μα πούν οι άλλε επιτροπέ που δεν έχουν στείλει προτάσει. Όμω να είστε βέβαιοι ότι ως το τέλος της διαδικασίας θα προσαρμόσουμε και τις τροπολογίες μας και τον ε, πίνακα με τα αριθμητικά στοιχεία για να προσπαθήσουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνοπτική εικόνα. Μεταξύ των απαιτήσεων, το όριο του 1,3 που δεν μπορούμε να πειράξουμε καθόλου και έπειτα των ε, τιμάτων που συχνά είναι θεμητά από τις επιμέρους επιτροπές για να προσαρμοστεί αναλόγως το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ιδού πρόεδρα η μέθοδος που ακολουθήσαμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Ζαμπέλ. Όλμπριχτ, Γιάνν Όλμπριχτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσθέσω απλώς όσα είπε η κυρία Τομά, ότι σε ό,τι φορά τον πίνακα με τα αριθμητικά στοιχεία, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τα αριθμητικά στοιχεία για καθένα από τα ερευνητικά προγράμματα. Δεν ήταν απλό, διότι η νέα ταξινόμηση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ίδια με την παλιά. Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα. Όταν εμείς ως Κοινοβούλιο ψηφίσαμε να προβελάξουμε και να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο η πολιτική συνοχή, το ερώτημα ήταν τι εννοούμε με αυτό. Εάν εννοούμε ότι το ERDF και το Κοινωνικό Ταμείο και τα Ταμεία Συνοχής πρέπει να παραμένουν στο ίδιο επίπεδο ή το νέο κεφάλαιο που λέει συνοχή και αξίες. Εννοούμε το Κοινωνικό Ταμείο ή το Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Οπότε, είπαμε ξεκάθαρα ότι όταν λέμε εννοούμε διατηρείται στο ίδιο επίπεδο, εννοούμε τα ίδια κονδύλια του ίδιου επίπεδου, όχι τα ίδια κεφάλαια, διότι τα κεφάλαια είναι άλλο πράγμα. Οπότε, οι επιμέρους επιτροπές υποχρεούνται να αναλύσουν μόνες τους ε, τα διάφορα επιμέρους αριθμητικά στοιχεία. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Διότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για τις διαφορετικές πολιτικές. Παράδειγμα, για το Ταμείο Συνοχής ε, σε σύγκριση με το Ταμείο Ανάπτυξης τη Επένθρου και το Κοινωνικό Ταμείο ή ένα εργαλείο της Αφέτει τα κονδύλια της Γεωργίας. Όλα αυτά είναι μπερδεμένα μεταξύ τους και περιμένουμε τις τελευταίες προτάσεις των ε, επιμέρους επιτροπών για την ε, ανάλυση των ε, αριθμητικών στοιχείων. Θα είναι μια σημαντική πολιτική ευθύνη των επιμέρους επιτροπών. Επίσης, η ενδιάμεση έκθεση δεν αφορά και δεν έχει να κάνει μόνο με τον πίνακα, διότι θα είναι απλώς ένα παράρτημα στην ενδιάμεση έκθεση. Ο Πίνακας αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο και ολόκληρη την επέτεια. Δηλαδή και τη διάρθρωση και τα ποσοστά και το πώς θα οργανωθεί το ε, Πουδουπού. Δηλαδή αν δεχτούμε τη νέα διάρθρωση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όχι. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο και επίσης έχει να κάνει και με την ευελιξία, την διαλεκτικότητα στο νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Η δουλειά μα λοιπόν είναι πολύ πιο μακρόπνοη από ότι τα σκέτα αριθμητικά στοιχεία. Όσοι εισηγητέ τη Επιτροπή Προπολογισμών ακολουθούμε όσα προέκυψαν από τα ψηφίσματα του Μαρτίου και του Μαΐου. Δηλαδή ότι εν γέννη για το που όταν λέμε 5 συν 5 θα πρέπει για πρώτη φορά να πούμε κατευθείαν 7. Αυτή είναι η πολιτική θέση του Κοινοβουλίου. Η διάρθρωση για μας μπορεί να είναι παραδεκτή, εννοείται, και η μείωση των προγραμμάτων που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι ως προς την ενδιάμεση αναθεώρηση. Από την προηγούμενη αναθεώρηση ε, και τη σχετική εμπειρία μας, θέλουμε να είμαστε σαφείς. Χρειάζεται πραγματική ενδιάμεση αναθεώρηση εδώ. Επίση, στην έκθεσή μα αναφέρουμε δύο στοιχεία. Ένα από αυτά αφορά τι δαπάνε και το άλλο θα το αναλάβουν οι εισηγητέ των ιδίων πόρων. Το κομμάτι για τους ίδιους πόρους, το έχουμε συμφωνήσει αυτό με την Ιζαμπέλ, ε, ακόμα το επεξεργαζόμαστε, γιατί και οι συνάδελφοι δεν έχουν ολοκληρώσει, αλλά έχει να κάνει και με το κράτο δικαίου αυτό. Το κράτος δικαίου είναι μια πολύ σημαντική ιδέα. Δεν θέλουμε να τα επαναλάβουμε όλα σε σχέση με τον νέο κανονισμό, αλλά αν ο νέος κανονισμός γίνει αποδεκτός από το Συμβούλιο και στη διαδικασία της συναπόφασης από το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία ότι δεν θα υπάρχουν τιμωρητικά μέτρα για τους τελικούς δικαιούχους, διότι το κράτος δικαίου και ό,τι αφορά το σύστημα της δικαιοσύνης, την λειτουργία του νομικού συστήματος, την πάταξη της διαφθοράς και το καθεξής, αφορούν και είναι θέμα ε, κυβερνητικής πολιτικής. Οι τελικοί δικαιούχοι δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν για κάτι που οι πολίτες δηλαδή να τιμωρηθούν για αποφάσεις που πήραν οι κυβερνήσεις τους. Είναι ένα κεφάλαιο αυτό. Συνοψίζοντα λοιπόν, η ενδιάμεση έκθεση θα είναι η πολιτική μα θέση. Η θέση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα του Πουδουπού. Ε, δηλαδή, με προτάσεις για τη διάρθρωση, με προτάσεις για την ευελιξία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και στοιχεία που είναι καινούργια, αυτά που ανέφερε η Ζαμπέλ. δηλαδή πρώτα απ' όλα τροπολογίες επί ακόμη και αν απλώ έχουμε το δικαίωμα τη συνένεση και τον πίνακα, ο οποίο θα είναι μια πάρα πολύ σαφή δήλωση του Κοινοβουλίου. Πώ κατανοεί δηλαδή το Κοινοβούλιο τη θέση του ανώτατου ορίου του 1,3%. Πώς μπορεί να αναλυθεί και να διαιρεθεί αυτό το 1,3%. Να θυμίσω, συναδελφοί, ότι αυτή τη στιγμή δεχτεί το σχέδιο της έκθεσης η Επιτροπή Προπολογισμών και ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο ενδιάμεση έκθεση. Στη συνέχεια, οι επιμέρους επιτροπές θα αναλάβουν να ψηφίσουν το νομοθετικό κείμενο που θα συμπεριλαμβάνει τους αριθμούς, τα αριθμητικά στοιχεία της ενδιάμεσης έκθεσης. Είναι σημαντικό αυτό γιατί πρόκειται για δύο παράλληλες οδούς, σαν να εργάζονται ταυτόχρονα δύο επιτροπές. Πρόεδρος, ευχαριστώ τους δύο συνεισηγητές μας για την ε, επιμέλεια που επέδειξαν στην επεξεργασία και τη σύνταξη αυτού του κειμένου, το χρόνο που αφιέρωσαν και τις πολλαπλές συνομιλίες που είχαν με συναδέλφους από άλλες επιτροπές. Για να είναι σε θέση για πρώτη φορά να υποβάλω μια πρόταση με ποσά αναπρόγραμμα. Κάτι που επιτρέπει να σχηματιστεί μια διαπραγματευτική θέση που μας διευκολύνει. Εφόσον βέβαια ισχύσει η θετική προοπτική ότι θα εγκριθεί η εντολή και από το Συμβούλιο και θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει στι αρχέ του 2019. Όμω το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο από μόνο το είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, αλλά συνδέεται και έχει και να κάνει πολλά με τη νέα ιδέα για τους νέους ιδίους πόρους. Εδώ έχουμε τέσσερις συνεισηγητές πέραν, από αυτούς που, πέραν αυτών που είναι υπεύθυνοι για, τους, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε και τους δύο που ασχολούνται με τους ίδιους πόρους. Ο κύριος Λεβαντόφσκι και ο κύριος Ντεπρέ πρώτη. Πρώτος, ο κύριος Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Μία, με μία φωνή μιλάνε οι δύο εισηγητές. Πολύ συχνά. Δεν είναι καινοτόμο η συνεισφορά μα σε αυτή τη ε, διάμεση έκθεση. Το μόνο που κάνουμε είναι να επαναλαμβάνουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το βασικό έχει ήδη αναφερθεί από τον Πρόεδρο. Σημείο 9. Για το single package δαπάνες και έσοδα ως ένα πακέτο. Δεν θα υπάρχει συμφωνία χωρίς αντίστοιχη προόδο για το νέο κεφάλαιο των ιδίων πόρων. Είναι η αιρεσιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει. Το σημαντικό για να μπορέσουμε να καθησυχάσουμε τον Ευρωπαίο πολίτη με το καθεστώς των νέων ίδιων πόρων είναι ότι οι νέοι ίδιοι πόροι δεν αυξάνουν το φορολογικό βάρος που φέρει στους ώμους του Ευρωπαίος πολίτη. Καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους νέους ίδιους πόρους που θα ευθυγραμμίζονται με την παγίωση και ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, τη φορολόγηση των εταιριών ε, των μεγάλων πολυεθνικών και την προστασία του περιβάλλοντος. Προσωπικός. Δεν καλυσορίζω και πάρα πολύ το θέμα των ίδιων πόρων και του ETS, του Trade Emission Scheme, ε, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχουμε μια σταδιακή εισαγωγή της ψηφιακής οικονομίας και να έχουμε και τον φόρο επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Όλα αυτά δηλαδή να είναι πηγές εισοδήματος για τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν να αποφέρουν. Και μαζί με τον Gérard Dupré εξετάζουμε τις επικοδομητικούς συμβιβασμούς και την επικοδομητική συνεισφορά στην όλη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, ο κύριος Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Γιάννης Λεβαντόφσκι εξέφρασε το ουσιώδες. Πολύ απλά θα ήθελα να σχολιάσω λίγο την επιλογή που κάναμε για μια σόφρονα θα έλεγα πολιτική προσέγγιση του θέματος. Να ευχαριστήσω και τους δύο άλλους συνεισηγητές γιατί ανάδειξαν τη σχέση που έχουν οι ίδιοι οι πόροι με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και πόσο άρρητα συνδεδεμένα είναι αυτά ε, στο επίπεδο της πολιτικής κακέρας και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, στη δήλωση σε ό,τι μας αφορά. Επομένως εμείς υιοθετήσαμε μια σόφρονα προσέγγιση με προσοχή, προσεκτική προσέγγιση γιατί, για δύο λόγους. Καταρχάς θέλησαμε να εντοπίσουμε τις αλλαγές στο σύστημα των ίδιων πόρων και να δούμε πού ακριβώς αλλάζουν τα πράγματα. Στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση και ο Γιάννου το ξέρει πολύ καλά και οι θέσει των κρατών μελών στη συζήτηση του Συμβουλίου αποκλίνουν τα μάλα. Δηλαδή, κρατημέλη δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα. Το σύστημα για αυτά τα κρατημέλη ε, των ίδιων Πόρων που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα είναι το α και το ω τελεία και παύλα. Για άλλα κράτη-μέλη όμως ε, η στάση τους είναι πολύ πιο ανοιχτή και στρέφονται προς την ιδέα να έχουμε νέους ίδιους πόρους από διαφορετικές πηγές στον προϋπολογισμό. Η συζήτηση είναι πολύ ζωντανή και πρέπει να ξέρουμε ότι σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους, το δικό μας κοινοβούλιο έχει λιγότερη εξουσία συγκριτικά με την εξουσία που έχει για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το κοινοβούλιο θα δώσει τη συγκατάθεσή του ή δεν θα τη δώσει. Ενώ για τους ίδιους πόρους δεν έχουμε λόγο. Μπορούμε να δώσουμε μια γνώμη, μια γνωμοδότηση, αλλά αυτά είναι λόγια του αέρα. Δεν υποχρεούνται στο Συμβούλιο να λάβουν υπόψη αυτό που λέμε εμείς για τους ίδιους πόρους και γι' αυτό συμφωνήσαμε. Να παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο τα πράγματα με προσεκτική στάση, δηλαδή να σταθούμε όσο δυνατόν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις προτάσεις της και να ε, προτείνουμε έτσι διακριτικά ε, κάποιες άγουσες, κάποιους νέους δρόμους που αξίζει τα κράτη-μέλη να βαδίσουν λίγο σε αυτά τα μονοπάτια, να δουν τι καρπούς θα φέρουν. Γι' αυτό διαλέξαμε αυτή την προσεκτική και σόφρονα στάση. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Είναι σαφές ότι οι νέοι ήδη οι πόροι δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αύξηση του φορολογικού άχθους για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Εάν υπάρξουν νέοι ήδη πόροι, αυτό που θα κάνουν είναι να ελαφρύνουν τους φόρους που επιβάλλονται σε εθνικό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μειωθεί η συνεισφορά των κρατών μελών στον προϋπολογισμό ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ λοιπόν τους τέσσερις συνεισηγητές για το έργο αυτό που έχουν φέρει σε πέρας εδώ και σχεδόν δύο χρόνια με προσήλωση, με στόχο προσήλωση, με μια καλώς εννοούμενη ξέρω κεφαλιά την οποία καλωσορίζουμε και για την οποία τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε να τηρήσουν την ίδια στάση ε, επίμονη και προσεκτική στις συζητήσεις με το Συμβούλιο. Ο κύριος Φερναντές θα πάρει το λόγο για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για το επόμενο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Θέλω να ευχαριστήσω <clears throat> για τη δουλειά τους όλους τους συναδέλφους, ε, τους εισηγητές για όσα έκαναν, τους κοιόδης εισηγητές, και όσου ήταν ε, υπεύθυνοι από τι άλλε επιτροπέ, μπορούμε να πούμε στου πολίτε στους πολίτες τη Ευρωπαϊκή Ένωση το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο, πανέτοιμο για να διαπραγματευτεί. Ελπίζαμε και το Συμβούλιο να ήταν έτοιμο. Και το επιθυμούμε αυτό. Είναι ζωτική σημασία φέτο να προλάβουμε ε, να έχουμε τη θέση του Συμβουλίου πριν λήξει η θητεία μα. Είναι ζωτική σημασία. Είναι ζωτική σημασία να επιτευχθεί συμφωνία σε σχέση με το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο σε αυτήν τη θητεία. Και αυτό δεν είναι για να ωφεληθούν οι πολιτικές ομάδες που είναι συσπηρωμένες ως προς το θέμα αυτό είναι προ όφελο τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των πολιτών. Οι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον απαιτούν να έχουμε πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και εγκεκριμένο, ώστε τα προγράμματα και οι πολιτικέ μα να μπορέσουν να ξεκινήσουν να λειτουργούν τον Ιανουάριο του 2021. Η διακοπή οποιοδήποτε προγράμματο θα ήταν δραματική μαζί με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα προγράμματα πρέπει να εγκριθούν ε, μαζί με τους σχετικούς κανονισμούς. Και οι περικοπές θα πρέπει να είναι κάτι που θα σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Φανταστείτε ε, αν, διακόπταμε το Erasmus Συν ή αν υπήρχαν διακοπές στις πληρωμές των γεωργών. Τι θα σήμαινε αυτό εάν η πολιτική συνοχή, η κοινωνική πολιτική για τις δημόσιες επενδύσεις, για τις χώρες που έχουν 70% κρατικέ επενδύσει ε, δεν είχαν αυτά τα μέσα. Τι θα γίνει με τα δημοσιονομικά μέσα που διαθέτουμε στι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει. Τι θα γίνει αν υπήρχε διακοπή εκεί. Οι νομικέ αμφιβολίε και οι νομικοί ενδιασμοί που θα προέκυπταν εάν δεν είχαμε έτοιμο προπολογισμό και έπρεπε να ανατρέξουμε στο σύστημα των 12 ε, τιμωρίων η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, είναι αξιόπιστη για τους επενδυτές και για τα ερευνητικά προγράμματα και την καινοτομία. Και αυτά χρειάζονται αξιοπιστία. Πρέπει να μπορούν να προβλέψουν οι άνθρωποι τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να τους αφήνουμε να σκεφτούν ότι θα υπάρξει διακοπή στα προγράμματα. Αυτό θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πλήξει την εδαφική συνοχή ε, και την αλληλεγγύη μας. Πρέπει να λύσουμε προβλήματα που είναι κοινά για όλου. Και είναι ζωτική σημασία η αλληλεγγύη και αυτή να εκφραστεί στην πράξη και από όλου. Χρειάζεται εδώ υπευθυνότητα. Έχουμε κοινέ προκλήσει. Τα μεταναστευτικά κύματα, την ε, ε, άμυνα και την ε, ασφάλεια. Αυτά απαιτούν κοινέ αποκρίσει. Αποκρίσει στην κλίμακα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ω προ αυτό και μάλιστα αυτά απαιτούν από εμά και οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το Συμβούλιο τι κάνει πρέπει να αναθέσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπραγματευτεί, ε, όπω και το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικότατα όλα αυτά για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη που μα αποδίδουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Ε, που, μας, ε, που θα πρέπει να μας αποδίδουν και που θέλουμε να, όπως ήδη συμβαίνει, να συνεχίσουν. Η πρότασή μας είναι το 1,3 του, του ΑΕΠ. Ε, είναι δικαιολογημένο αυτό. Η μέθοδος που ακολουθούμε στο Κοινοβούλιο είναι απλή και bottom-up. Είναι λογική. Ε, έχουμε για κάθε πρόγραμμα, για κάθε πολιτική συγκεκριμένα ποσά αυτά που απαιτούνται. Ε, ας κάνουμε τους λογαριασμούς και ας βρούμε τι χρειάζεται. Δεν είναι τίποτα φοβερό αυτό που ζητάμε από το ΑΕΠ των ε, μελών. και έτσι διατηρούμε και τη συνοχή, τη γεωργία, ενισχύουμε την έρευνα, ε, στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, προσαρμόζουμε το Erasmus Συν ε, με αυτό είμαστε σε θέση να ε, υποστηρίξουμε την ε, άμυνα και την ασφάλεια, την τεχνολογική μας ανάπτυξη. Μερικοί θέλουν να έχουμε ένα ποσοστό, γενικό και αόριστο, αόριστο γενικό και αόριστο όριο, και μετά ανάλογα με τι προτεραιότητε να το προσαρμόζουμε. Όχι, για τι προτεραιότητε των Ευρωπαίων Πολιτών δεν μπορεί να γίνει έτσι. Ω προ τη χρηματοδότηση, υπάρχει ένα σημείο που είναι καθοριστικό και θα πρέπει να αποσαφινιστεί. Δεν έχουμε ευρωπαϊκούς φόρους. Ε, είναι αρμοδιότητες οι φόροι των ε, εθνικών κοινοβουλίων. Πώς θα έχουμε λοιπόν ε, εισοδήματα, έσοδα, χωρίς να βαρύνουμε τους φορολογουμένους. Γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσει και συζήτηση για τους ιδίους πόρους ακόμη και αν βρίσκεται κυρίως στα χέρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όμως, δική μας δουλειά και πρόταση των εισηγητών είναι να κάνουμε μια θετική πρόταση για να μειωθούν οι αντισταθμίσεις, να σταματήσουν οι εκτόσεις και τα rebate, να μετατραπεί ο προϋπολογισμός σε κάτι που θα έχει διαφανέστερη διάρθρωση. γιατί έτσι θα είναι σαφέστερο πώς ε, πρεκοδοτείται αυτό ο προπολογισμό και θα είναι και σαφή αυτά που θα πούν οι συγητές. Αυτά για να μπορέσει το Κοινοβουλίο να επιδιώξει αυτόν τον πολύ συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή ένα προπολογισμό στο ύψο των προκλήσεων και των δυσκολιών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που ανταποκρίνεται στι απαιτήσει των πολιτών και που επιτρέπει τον Γενάρη να ξεκινήσουν να λειτουργούν κανονικά όλα τα προγράμματα. Ευχαριστούμε. Μακάρι να σας ακούσει και το Συμβούλιο. Η Έντερ, ο Γκαρδία Θάμπαλ. Μα είναι και ο Βιώτη εδώ, που είναι ο Σκιώδης. Α, ναι, κύριε Βιώτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους τέσσερις συνεισηγητές, διότι πραγματικά η δουλειά που κάνουν και σε σχέση με όσα του ζητήθηκαν και τις θέσει τη Επιτροπής αυτή μετά από μήνες συζητήσεων είναι θαυμάσια. Θέλω να επικεντρωθώ στο τμήμα που είναι της δικής μας αρμοδιότητας, διότι η κυρία Τόμα ήδη παρουσίασε τις βασικές ιδέες για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ ήθελα λοιπόν να μιλήσω κυρίως για τους ιδίους πόρους. Πώς μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τον προπολογισμό. Και σε σχέση με όσα είπαν οι δύο συνεισηγητές, ακόμη και αν ξεκινήσαμε με μια σχετική ένταση, ε, προλαμβάνοντας ε, το πώς θα συζητηθούν στο επίπεδο των ιδίων πόρων, Σωστά τα είπαν ε, και ο κύριος Ντεπρέ και ο κύριος Λεβαντόφσκι. Χρειάζεται ρεαλισμός περισσότερο από πάθος. Δηλαδή σε σχέση με, τον, ε, με την επιθυμία του Κοινοβουλίου να υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα και όσα ζητήσει ίσως να ξεπερνούν τις προσδοκίες των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων. Πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν σε μερικά μέτρα ε, προγράμματα προτεραιότητας που να μπορούν όμως και ρεαλιστικά να γίνουν αποδεκτά από το Συμβούλιο και τελικά να εγκριθούν εάν το θέλει το Συμβούλιο. Αυτή νομίζω είναι η καλύτερη οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Το λέμε από την αρχή και με ενδιαφέρει πολύ και μένα και το άκουσα να το λέει και ο κύριος Λεβαντόφσκι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που ε, πήραν το λόγο μετά. Με ενδιαφέρει λοιπόν πολύ να είναι σαφές, απολύτως ξεκάθαρο, ε, για τα κράτη-μέλη, ακόμη και αν δεν είναι απόλυτα προετοιμασμένα, αλλά και για του πολίτε να είναι σαφέ ότι το δικό μα θεσμικό όργανο, το Κοινοβούλιο, δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να ε, επιβάλλει περισσότερου φόρου στου Ευρωπαίου πολίτε. Έχει απλώ την πρόθεση να εντοπίσει για να τροφοδοτήσει προγράμματα τα οποία είναι χρήσιμα και επικοδομητικά για τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν πετύχει, ε, έχουν ήδη δείξει την επιτυχία τους και θα συνεχίσουν να τη δείχνουν και να απελευθερώσουμε και πόρου για τα κράτη-μέλη που κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ο στόχο είναι να εντοπίσουμε πόρου πόρους ε, που να μην ε, είναι κάτι που θα βαρύνει τους πολίτες αλλά που θα χρηματοδοτήσει τα προγράμματά μας, όλο αυτό θα επιτρέψει και στα κάτι μέλη να έχουν περισσότερα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Το Κοινοβούλιο πάντοτε τέτοιο στόχο είχε. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Όπως είπατε κι εσείς, είναι αξεδιάλυτη η σχέση των δύο αυτών θεμάτων. Ακόμη και αν οι αρμοδιότητε του Ευρωκοινοβουλίου είναι διαφορετικέ ε, για του ιδίου πόρου και το πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι λοιπόν εντελώ αλληλένδετα τα δύο αυτά πράγματα. Το πού πού και ήδη οι πόροι που θα διαμορφωθούν τα επόμενα χρόνια ο σύστημα. Ευχαριστώ. Merci, monsieur. Σας ευχαριστούμε και εσά, κύριε Βιώτη. Εκπροσωπήσετε και την ομάδα Σοσιαλιστών Δημοκρατών για το ECR, κύριο Κέλμελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τους συνεισηγητές ε, για την πολύ καλή τους ε, ευσυνείδητη δουλειά. Ξέρουμε πόσο ε, πολλή δουλειά συνεπάγεται όλο αυτό. Οι θέσεις του Κοινοβουλίου ήδη είναι σαφής μέσα από διάφορα ψηφίσματα. Καλό είναι πάντως για μια ακόμη φορά να πούμε ότι εμείς ως ECR έχουμε διαφορετική άποψη σε πολλά θέματα, ιδίω ό,τι αφορά το πώς μπορεί να καταρτιστεί ένας αποτελεσματικός ευρωπαϊκός προπολισμό. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία. Έχουμε ακόμη την, ευκαιρία και την τύχη, θα έλεγα, με βάση τον, τα ψηφίσματα που έχουμε, να έχουμε ε, με τα διάφορα θέματα ε, εξηγήσει πολύ ξεκάθαρα το τι θέλουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλές φορές ε, χρειάζεται, ε, θέλουν κάποιοι περισσότερη ανακατανομή ε, των ήδη φυστάμενων κονδυλίων. Εμείς θέλουμε περισσότερα. Λέμε ότι έχουμε νέες προκλήσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι όμως άπειρο το χρήμα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε τολμηροί. Πρέπει να προτείνουμε, παραδείγματο χάρη, και να προβλέψουμε για τη γεωργία μείωση των κονδυλίων. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα επταετή προ προγραμματισμό και να προβλέπουμε και για τα 7 έτη τα ίδια ποσά και μετά ε, να ξανατεθούμε ενώπιον του διλήμματος μετά από την επταετία ότι ε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα εντελώς γιατί βασίστηκαν πολύ σε αυτό και ξαφνικά να φτάσουμε στο ιωρικό τομέα και να πούμε ότι πρέπει να γίνει μια ανακατανομή των κονδύλων, να διατεθούν αλλού. Ε, περνάω στην πολιτική συνοχή. Φυσικά και μπορούμε να δείξουμε αλληλεγγύη, αλλά ε, την πολιτική συνοχή δεν τη χρειαζόμαστε για τις περιφέρειες που ε, είναι πάνω από το μεσόρο. Δεν τις χρειάζονται, δεν χρειάζονται αυτά τα κονδύλια αυτές οι περιφέρειες. Θέλουμε για αυτές τις περιφέρειες που τη χρειάζονται τη συνοχή να διαθέσουμε τα κονδύλια. Και εκεί πρέπει να είμαστε τολμηροί και να βρούμε, να εισαγάγουμε μία μέθοδο με την οποία θα ορίσουμε στόχους και τους οποίους θα μπορούμε να μετρήσουμε. Γιατί δεν είναι δυνατόν να περιγράφουμε κάτι επί χάρτου... και τελικά κανένας να μην ενδιαφέρεται στην πράξη για το πώς αυτό επετεύχθη στην πράξη με τα χρήματα, με τους πόρους. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους, και εκεί έχουμε διαφορετική άποψη σε σχέση με αυτά που άκουσα εγώ σήμερα. Και πραγματικά κάπως με εκπλήσει αυτή η εκτίμηση, σχεδόν μάντρα και αρχές και αξιώματα αναφέρουμε εδώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σίγουροι εντελώς ότι το σύστημα αυτό δεν θα επιβάρει περισσότερο τους Ευρωπαίους πολίτες. Τι συνάδελφοι, θα ήθελα σας παρακαλέσω να δείτε την ιστορία ε, και στα κράτη-μέλη μήπως υπήρχαν μεγάλοι τομείς όπου επειδή υπήρξε ε, ένας φόρος ο οποίος ε, εισήχθη να δημιουργήθηκαν εκεί άλλα προβλήματα. Δηλαδή όταν έχουμε ένα φορολογικό δίκαιο αυτό έχει να κάνει και με μάλλον δεν έχει καμία σχέση με το πώς εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. και πολλές φορές δεν θα μειωθούν οι φόροι στα εθνικά κράτη, με αποτέλεσμα πρέπει οι πολίτες να βαρεθούν ακόμη περισσότερο. Επίσης, αν θέλουμε ε, μια αλληλέγγυα Ευρώπη, δεν χρειάζεται φορολογικό δίκαιο, ε, γιατί ε, αν χρειάζεται κανείς ε, απόδειξη για κάτι τέτοιο, ας πάει να δημιουργήσει Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, μάλλον Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης ή κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεπρέ τώρα για την ομάδα Άλντε. Ευχαριστώ. Θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον κύριο Τόρβαλτ. Ωστόσο, ένα δευτερόλεπτο να αντιδράσω σε αυτά που είπε ο συνάλφος Κέλμελ. Όταν μιλάμε για νέους ίδιους πόρους, κύριε Κέλμελ, δεν μιλάμε για ευρωπαϊκούς φόρους, για ευρωπαϊκό φόρο, παραμένουν εθνικοί οι φόροι, αποφασίζονται αυτοί οι φόροι από τους υπουργού. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου πρέπει να, τις ψηφι... να τους ψηφίσουν τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και ένα μέρος μόνο των εσόδων αυτών μπορεί ε, να ε, διατεθεί στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Μην κυνηγάτε φαντάσματα. Μάλλον εμείς πρέπει να κυνηγήσουμε αυτό το φάντασμα του Ευρωπαϊκού Φόρου που αφήσατε να ε, πλανάτε, κύριε Κέλμελ. Να είμαστε ξεκάθαροι. Τώρα, στόχο των δύο πόρων ποιος είναι να μειωθούν σύν το χρόνο των κρατών μελών που επιβαρύνουν τον εθνικό προπολογισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό ήδη το βλέπουμε γιατί σε σχέση με την κατάσταση που γνωρίσαμε κατά το παρελθόν το μερίδιο των ιδίων πόρων που βασίζεται στο εθνικό εισόδημα και καταλογίζεται στον εθνικό προπολογισμό μειώνεται στο πλαίσιο τη προκοδότησης του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Θα το πω αυτό με κάθε, ε, με όλα τα φιλικά αισθήματα που τρέφω προς εσά, Κύριε Κέλμελ. δεν ζητούμε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού ε, Φόρου. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στον, αν συμφωνείτε βέβαια, στον συνάδελφο. Εγώ θα του δώσω το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Τέλος πάντων, με άλλα λόγια, αυτή οι νέοι διποροί είναι φόροι. Α, και οι τελωνιακοί δεσμοί εισπράττονται από τα κράτη-μέλη. Βεβαίω, βεβαίω, λέει ο κ. Δεπέρα, τα κράτη-μέλη. πρόεδρο, που διατηρούν το 20% με την κατάσταση. Ε, αυτό θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε, αλλά τέλο πάντων κρατάνε το 20% για τι δικέ του ανάγκε. Άμστερνταμ, Ρότερνταμ και Αμβέρσα. Λοιπόν, κάποια στιγμή, δεν ξέρω, πρέπει να δούμε μήπως είναι 20%, το 20% αυτό για τις ανάγκες Βελγίου και Λανδίας πως είναι πολύ ε, ως ποσοστό. Αλλά οι διπόροι είναι φόροι οι οποίοι θα εισπράττονται. Υποθέτω ότι οι εθνικές νομοθεσίες θα προσαρμοστούν ως προς αυτό και θα εισπράττουν τα κράτη-μέλη και θα διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα να μειωθεί η εισφορά των κρατών στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και αυτό κύριε Κέλμερ θα επιτρέψει να μειώσουν τους άλλους φόρους που επιβάλλουν στους φορολογουμένους στα κράτη-μέλη. δεν θα επιβαρύνουν ήδη οι πόροι το φορολογικό άχθος των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Κύριε Τόρβαλτς, τώρα έχετε εσεί το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ε, εκ μέρου ε, του Νίλς, ε, μιλώντας ως ένα κορίτσι, ως μια απλή Ευρωπαία πολίτης. Γιατί οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν άμεσα εκατομμύρια κορίτσια. Γι' αυτό και θα ήθελα στην, στην εισαγωγική μου παρέμβαση να πω ότι εμείς τα κορίτσια αυτό που ζητούμε είναι μια ε, απάντηση. Ε, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί ε, σε αυτό που ζητούμε. Θέλουμε έναν προπολογισμό υπεύθυνο που να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φίλου να επενδύει στα κορίτσια, στο μέλλον μα, στην αντιμετώπιση των διακρίσεων, διότι η ισότητα των φίλων δεν είναι λόγια μόνο που τα λέμε δεξιά και αριστερά, αλλά είναι κάτι αναγκαίο για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για την ποιότητα της ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Αν θέλουμε όλοι αυτοί να ζουν ωραία και καλά. Εμείς ε, θέλουμε να μας ακούσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμάς τους νεαρούς σε ηλικία πολίτες. Θέλουμε ένα πολιτές μας πλαίσιο το οποίο να αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα τις αξίες που θέλουμε και να τα αποκρίνεται στις υποσχέσεις που μας έχουν γίνει με όλες αυτές τις πολύ ωραίες ομιλίες που έχουμε ακούσει. Δεν θέλω να νιώσεις, ε, Νίλης, τελείως ε, άχρηστος. Θα σου δώσω το σολόγο να πεις και εσύ δύο λόγια για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Thank you, thank you, And when her first name, I think... Ευχαριστώ πολύ. Αν κάνετε ένα διάλειμμα από το προϋπολογισμό, ε, διαβάστε εθνικό ποίημα Κάλαβαλα, που το πρώτο, το μικρό το όνομα της... Ε, Άινου αναφέρεται. Τέλο πάντων, ε, δεν θέλω να μιλήσω για σοβινιστικά γουρούνια, είναι ένα φιλανδικό τέλο πάντων ε, θέμα το οποίο επανέρχεται. Θέλω να ευχαριστήσω του ε, συνεισηγητέ για τη σκληρή του δουλειά που δεν έχει τελειώσει και στο μέλλον έχουν να, να κάνουν πολλά μέχρι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα μιλήσω πιο πολύ από το πρίσμα και της δημοσιοποίησης της έκθεσης της IPCC, της ε, Επιτροπής για το Κλίμα, που δημοσιοποιήθηκε χθε η έκθεση αυτή. Η ενδιάμεση αναδρόση, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει μεγάλη σχέση με το κλίμα. Διότι αν δείτε, φαντάζομαι έχετε ήδη δει κάποια από τα χθεσινά νούμερα, αν δείτε την καμπύλη αν δεν μπούμε εντό ε, της καμπύλης με τις σημερινές μας αποφάσεις, τότε θα χάσουμε το τρένο. Και επομένω, πανερχόμενο στην διάμεση εξολόγηση και ακούγοντας ε, και τις ε, επιθυμίε, Άινο, έχουμε πραγματικά δουλειά μπροστά μας. Με στόχο ε, να πάρουμε αποφάσεις που ξέρουμε ότι θα επηρεάσουν όχι τόσο τις δικές μας, αλλά τη δική της ζωή στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Η ευθύνη των ανδρών δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη όσο είναι σήμερα. Γιατί με τις δικές μας ε, υπερβολές ανδρών και γυναικών μπορούν να κάνουμε πραγματικά τη ζωή ανυπόφορη σε αυτό τον πλανήτη και αυτό είναι πολύ δυστυχές. Ο κύριος Σολέγη από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και τους συνεισηγητές για τη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι αυτού του σημείου. Είναι μια πολύ καινοτόμο προσέγγιση αυτή που έχουν υιοθετήσει με την έκθεση αυτή. Κυρίως χάρη στο δεύτερο μέρος με τις νομοθετικές τροπολογίες και με το τρίτο μέρος με την ε, ανάλυση σε αριθμούς και ψηφία. Θεωρούμε την έκθεση ιδιαίτερως ευπρόσδεκτη, γιατί αντιπροσωπεύει και εκφράζει τις προηγούμενες θέσεις που έχει οθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση του Μαρτίου και στο ψήφισμα του Μαΐου. Θεωρούμε ότι το σχέδιο έκθεση συμφωνεί με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε έτοιμοι να παραμείνουμε στο ίδιο στρατόπεδο, να ψηφίσουμε με τον ίδιο τρόπο όπως ψηφίσαμε και πριν. Θα θέλαμε όμως ορισμένες βελτιώσεις στο κείμενο. Μετά από συζητήσεις και που θα έχουμε. Και θα ήθελα να τονίσω κάποια σημεία σημαντικά για την ομάδα μας για τους ε, ε, ε, στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χιλιετίας, τα θέματα του φύλου, όλα αυτά είναι προτεραιότητες για μας. Πράγματι υπάρχουν στο σχέδιο κειμένου, αλλά πρέπει να βελτιωθεί το κείμενο ως προς αυτή τη διατύπωση στα δύο πρώτα τμήματα της έκθεσης. Πιστεύουμε ότι η έκθεση θα πρέπει να αποφαίνεται για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε ο στόχος το 25% των δαπανών να γίνεται και να διοχετεύεται έτσι ώστε να συμβάλλει στην καταπολέμηση ε, της κλιματικής αλλαγής. Εμείς προτείναμε 30% δαπάνες να σχετίζονται με το κλίμα το συντομότερο δυνατό, το αργότερο μέχρι το 2027. Θα πρέπει να βρεθεί μια συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα διατυπωθούν αυτές οι συμβιβαστικές λύσεις. Ο προπολογισμό στο νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι πιο πολύ στραμμένο στα θέματα του φύλου, που θα πρέπει να βρίσκονται σε όλες τις ε, επικεφαλίδες και σε όλους τους τίτλους να μην αποκλείουμε επιλογές στην ενδιάμεση αναθεώρηση, η οποία οφείλει να είναι ευκαιρία για αναθεώρηση και πραγματικά βελτίωση. Το ίδιο ισχύει για όλο το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ούτως ή άλλως και αν χρειαστεί να ανανεωθεί και να μεταρρυθμιστεί και σε βάθος μάλιστα. Είμαστε υπέρ με των αυξήσεων του προϋπολογισμού σε ορισμένα προγράμματα. Θα αναφερθώ σε ένα μόνο το ESF+, το ESF SIN και τα νούμερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μείωση, σημαίνει μείωση. Εμείς προτείνουμε ελαφρά αύξηση, αλλά όχι και τεράστια μείωση όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να σεβαστούμε τα συνολικά κατόφλια του 1,3% όπως αναφέρονται στην έκθεση του Μαρτίου να υπενθυμίσουμε την πάγια μας θέση ότι ο κανονισμός για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να υιοθετείται με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε τη διατύπωση που θα έλεγε ότι σε κάθε περίπτωση το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να εγκρίνεται πριν από τις εκλογές. Δεν αποκλείουμε την πιθανότητα να εγκριθεί πριν από τις εκλογές, ωστόσο για εμάς το περιεχόμενο είναι πολύ πιο σημαντικό από το χρονικό όριο και τη χρονική προθεσμία. Άρα η θέση και η, η ψήφος μας θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο των προτάσεων που θα ε, προκύψουν από το Συμβούλιο. Και για τους ίδιους πόρους θα ήθελα να πω δύο λόγια. Πρώτον, Θεωρούμε ότι το κείμενο πρέπει να ενισχυθεί και να είναι πιο κατηγορηματική η διατύπωση, ειδικότερα για το CCCTV, το EFTD και το ψηφιακό φόρο. Με αυτά τα στοιχεία θα πρέπει όλα αυτά να είναι πιο ισχυρά και συμφωνούμε με τη θέση του Κοινοβουλίου για τις εκπτώσεις και δεν συμφωνούμε με την πρόταση phasing out σταδιακής εξάλληψης γιατί αυτός είναι ένας τρόπος να παραταθεί τελικά επαόριστον κάτι που σαφέστατα είναι ανομαλία. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες σχετικά που λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις που έκανα μόλις τώρα. Και βεβαίως ευχαρίστως να συνεργαστούμε και με τους εισηγητές και τους υπολείπους για την ε, ε, βελτίωση του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω για την ΚΟΕ να είναι κανείς εδώ. Ο κύριος Βαλή από το EFTT. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για τις ε, εισηγήσεις τους, αλλά δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ότι όταν κάποιοι λένε ότι μερικά προγράμματα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Συμφωνώ απολύτω με την καταπολέμηση τη φτώχεια, τα κονδύλια για την έρευνα. Συμφωνώ και με τον συνάδελφο Τόρβαλτ που ζητά κονδύλια για προγράμματα που εξυπηρετούν και ωφελούν του νέου. Όμω θα πρέπει να είμαστε και και να αποφύγουμε να γινόμαστε λαϊκιστές διότι και εγώ μπορώ να σκεφτώ πολλούς σεισμοπαθείς από την κεντρική Ιταλία και θα μπορούσα να αρχίσω να μιλάω για όλα αυτά τα προβλήματα και το τι πρέπει να γίνει με τις δαπάνες και κυρίως σε κρατικά κονδύλια που δεν επιτρέπουν την ανοικοδόμηση και που υπάρχουν ζημιές ας πούμε και αυτά είναι περιορισμοί που έρχονται από την, ε, ε τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για 100 δις στη χώρα μου κόστος. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε τι συμβαίνει σήμερα, να δούμε τι θα συμβεί και με το Brexit και να αποφύγουμε να κάνουμε προτάσεις που μπορεί να είναι υπέρμετρα ε, μη ρεαλιστικές. Εάν βρεθούν επιπλέον πόροι, προφανώς και θα είναι και πάνω, περισσότερο από υποφερτό θα μπορούσε να υπάρξει συνεισφορά δεκάδων δις παραπάνω. Δεν ξέρω αν τώρα η αυστηρότητα και η λιτότητα και όλοι αυτοί οι περιορισμοί του προπολογισμού επιτρέπουν τέτοιου είδου τροφοδότηση αυξητική. Ωραία λοιπόν ακούγονται όλα αυτά, αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο να επιτευχθούν. Και από τη δική μου τη σκοπιά θα ήθελα να γίνει μια δουλειά πολύ περισσότερο σχολαστική, στο να προσπαθήσουμε να δούμε πού υπάρχουν ε, περιττές δαπάνες στο επίπεδο του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Θα πρέπει να γίνει κάποια μετακύληση κονδυλίων σε προγράμματα που θεωρούμε ότι είναι αναπηρκή ή να δούμε τι άλλα προγράμματα έχουν πραγματικά ε, αρνητικές επιπτώσεις ε, ως προς την χρήση των κονδυλίων. Ξέρω εγώ η Τουρκία που βλέπουμε ότι είναι μια χώρα με πολλά προβλήματα και τα κονδύλια που παίρνει είναι τρεις γραμμές που θα μπορούσαμε ήδη να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε πώς θα δώσουμε περισσότερα κονδύλια σε άλλα προγράμματα. Και κάτι σημαντικό που θα ήθελα να γίνει κατανοητό και θα το συζητήσω μετά και με του υπόλοιπου συζητητέ για να φωτίσουμε το θέμα, είναι τα rebate, οι ε, δηλαδή. Δεν ξέρω αν τέτοιου είδου εκτόσεις είναι ε, ε, ωφέλιμες πλέον ε, στον πεδίο του προπολογισμού και υπάρχουν τόσα πολλά rebate στον προπολογισμό μας που κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε. Δεν μιλάω μόνο για το. Για την έκπτωση αυτή, την επιστροφή τη Αγγλίας που λόγω του Brexit θα πάψει να υπάρχει. Αλλά υπάρχουν και άλλε χώρε άλλες χώρες που έχουν τέτοιου είδου έκπτωση. Αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσουμε και να δούμε πώς θα χειριστούμε την κατάσταση στο μέλλον. Πάντως θα τα συζητήσουμε και στο μέλλον με τους συναδέλφου και ελπίζω ότι θα επιστρέψουμε στην πραγματικότητα των αριθμών χωρίς να κάνουμε τίματα που μπορεί να θεωρηθούν και υπέρμετρα λαϊκιστικά. Par la voix de leur coordinateur. Ε, ευχαριστούμε. Όλε οι πολιτικέ ομάδε εκφράστηκαν μέσω των εισηγητών και των εισηγητών του. Τώρα θα δώσω το λόγο στου υπόλοιπου συναδέλφου. Ο πρώτο είναι ο κύριο Μάνκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω από τη μια πλευρά ότι πολλά κράτη-μέλη ε, θεωρούν ε, τα, τις εισφορές ως μεταφορές πιστώσεων και όχι τόσο ως επενδύσεις. Εμείς είχαμε βρει ε, και κατά το παρελθόν μια λύση για τους ίδιους πόρους, η οποία δεν πέρασε γιατί κάποια κράτη, κάποιες κυβερνήσεις θεώρησαν ότι δεν θα είχαν πλέον καμία ευθύνη. Όμως αυτό είναι λάθος. Δεν θα είχε αποδυναμωθεί η θέση των κρατών μελών, δεν θα είχε αποδυναμωθεί το Συμβούλιο. Έγινε τέλο πάντων αυτή η ομάδα, μπορούσαν να ορίσουν τα κράτη τρεις εκπροσώπους ε, και καταλήξαμε σε μια πρόταση η οποία τέλος πάντων δεν έγινε τελικά ε, δεκτή. Ε, Είχα ζητήσει να μας πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έγινε ε, με το φόρο άνθρακα, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να βοηθήσει στη χρηματοδότηση του επτάετους προπολογισμού. Θα το λάβουν υπόψη επί Κομισιό. Γιατί τελικά όμως δεν ελήφθη υπόψη, ενώ είπαν θα το λάμβαναν υπόψη. Τι να τον κάνουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αν δεν είναι προφανές για τον ευρωπαίο πολίτη. Ε, και μετά έχουμε νέα Brexit και στο μέλλον. πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάνω απ' όλα την ευεξία, την ευημερία μάλλον των πολιτών. Τώρα για το να νάθρακα πράγματι, αυτά που έγιναν θα έπρεπε ίσως να τα ξαναδούμε. Κύριε Κρέσλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ερωτήσεις. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτή η εγγύηση για τα παιδιά ακριβώς, αυτό το child guarantee. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι. Επίσης, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Πραγματικά, αν ε, υπάρχει αυτή η πρόταση και αν μιλάμε τώρα για το κράτος δικαίου, λέμε ότι θα έχει δημοσιονομικές ε, συνέπειε, αλλά όχι για τους ε, δικαιούχε. Ε, πραγματικά δεν πρόκειται να δουλέψει αυτό και ότι σίγουρα πρέπει να είναι και θα είναι αισθητό αλλά μην αυταπατώμεθα τώρα για την τροπολογία αυτή το καταλαβαίνω ότι θέλουμε να παραμείνει το πρόγραμμα σε ισχύ και σε λειτουργία αλλά αν υπάρχουν προβλήματα με το κράτο δικαίου με μια χώρα οι αστυνομία, η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί. Αυτό σημαίνει. Επομένως ε, ε, υπάρχουν προβλήματα και με τους δικαιούχου Θέλω να αναφέρω την περίπτωση της Ουγγαρία που έχουμε τελικό δικαιούχο ε, που δημιουργήθηκε με αυτόν πρόβλημα και δεν μπορούμε να εργαστούμε με την εθνική δικαιοσύνη στην προκειμένη περίπτωση. Επομένω, δεν οδηγεί πουθενά, νομίζω, αυτό ο στόχο. Και νομίζω ότι η Κομισιόν έκανε μια καλή πρόταση. Σε ό,τι αφορά τώρα τι τροπολογίε ε, για την ε, ε, το Ευρωζώνη, έχουν διαγραφεί. Πώς τη βγάζουμε από το κράτος δικαίου και την τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης. Είναι λάθος. Ε. Είναι σημαντικό ε, να τηρείται το δίκαιο στην Ευρωζώνη, γιατί αν δεν γίνεται αυτό καταραίει, ε, διασπάται η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά. Ξέρω τι πρέπει να γίνει. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλή και στρέφεται προς το σωστό στόχο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν το καταλαβαίνω ότι σκοπό είχε αυτή η τροπολογία. Νομίζω ότι η Κομισιόν έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση. Ό,τι αφορά ε, να μπει στον προπολογισμό του Ταμείου είναι καλό, αλλά τα άλλα δύο πραγματικά έχω δυσκολίε για τα άλλα δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκρέσλε. Έχουμε κοινή συναδρίαση, Κοντ Μπάτζ αύριο το μεσημέρι. Ακριβώς ε, με θέμα τους κανόνες που έχουν να κάνουν με το σεβασμό του κράτους δικαίου. Το, λόγο έχει ο κύριος Σαρβάμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω τρία ε, θέματα που θα ήθελα να σας αναφέρω. Καταρχάς να συγχαρώ τους εισηγητές και τους συνεισηγητές ε, για την πολύ σκληρή δουλειά τους, για τις προτεραιότητες. Συνεχώς ε, προσπαθούμε να τα εξισορροπήσουμε όλα αυτά και να ε, έχουμε όλα τα μπαλάκια στον αέρα σαν να επιδέξει ακροβάτες και για τη γεωργία και για τη συνοχή και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για το κλίμα και για το μετανάστευση και για το ένα και για το άλλο. Ε, αν θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, ακόμα και με το 1,3% που είναι ο στόχος μας, πάλι δεν θα φτάσει για να ε, προχωρήσουμε όλες μας τις προτεραιότητες. Επομένως, ε, τι θέλω να πω με όλα αυτά. Να είμαστε ξεκάθαροι για το ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Όποιες και αν είναι, δεν τις κρίνω, ούτε θα τις απαριθμίσω με σειρά ιεραρχίας. Όμως, αν ρωτήσουμε τον Ευρωπαίο πολίτη, και τον έχουμε ρωτήσει, είναι πολύ σαφές τι πιστεύει ο Ευρωπαίος πολίτης ότι ε, είναι η προτεραιότητα. Πρώτον, ασφάλεια. Δεύτερον, μετανάστευση. Τρίτον, κλίμα κλιματική αλλαγή. Ίσως αυτά πρέπει να δουλέψουμε. Ε, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω εγώ να υπογραμμίσω ως σαφές την προτεραιότητα που δεν υπάρχει ακόμα είναι το safe και η μεταφορά. Οι μεταφορές. Είναι ο φτωχοδιάβολος, ο κακομύρης, ο ξεχασμένος που κάθε κράτος μέλος τον ε, παραπετά. Και ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο. Όμω εκεί σε αυτό το πεδίο μπορούμε εμεί να ακομίσουμε πραγματικά προστιθέμενη αξία. Άρα να διαχωρίσουμε ξεκάθαρα ποιε είναι οι προτεραιότητές μας. Και δεύτερο, ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Είναι μια τελείω διαφορετική διάσταση στο εγχείρημα αυτό που προσδίδουμε. Δεν είναι τόσο και μόνο επί της ουσίας. Είναι η στοχοπροσύλωση στα αποτελέσματα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό τον προορισμό σε γενικές γραμμές δεν είμαστε ακόμα ξεκάθαροι. Και δεν λέω ότι η αδιάμεση έκθεση πρέπει να είναι υπερβολικά ξεκάθαρη. Λέω ότι αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κείμενο. Δηλαδή, τα χρήματα του φορολογουμένου να τα βάλουμε να δουλέψουν και να αποδώσουν. Περί αυτού πρόκειται. Να έχουμε σαφείς ορισμούς δηλαδή. Και τρίτον, το κράτος δικαίου. Είμαι συνδυσηγητής με την κυρία Καρτία Θαμπάλ για αυτό το θέμα και αξιοποιώ την ευκαιρία, δράτω με τις ευκαιρίες για να απευθυνθώ στην κυρία ε, Γκρέσλε και να της πω ότι το θέμα και το ερώτημα που θέσατε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι σαν να προσπαθούμε να τετραγωνίζουμε τον κύκλο. Δηλαδή, πώς γίνεται να κλείσουμε τα χρήματα και να μην τα δώσουμε, αλλά να μην επαρεαστούν οι τελικοί δικαιούχοι. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό, θα το σχολιάσω στη δική μου έκθεση για το κράτος δικαίου. Ωστόσο, στο τέλος, πρέπει να υπάρχει νόημα, πρέπει πραγματικά αυτό να βοηθά το κράτος δικαίου, να βοηθά έτσι ώστε να ε, αντιστραφεί η κατάσταση σε σχέση με το κράτος μέλος που δεν σέβεται το κράτος δικαίου. Στην ενδιάμεση έκθεση δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, ε, γιατί αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μπάγκιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα την χαρά να συνδεπραγματευτώ ε, τη, για το πολιτές πλαίσιο. Εντάξει, δεν ήταν πάντα χαρά. Ε, κάποιες φορές ε, ήταν και δύσκολο, αλλά χρειάζεται να μπορούμε να διαπραγματευτούμε ε, και σίγουρα θα πρέπει να μπορούμε να λογοδοτούμε και στους Ευρωπαίους πολίτες και έχοντας υπόψη το ε, ταχύως μεταβαλλόμενο κόσμο με τα μεγάλα προβλήματα, με την παγκοσμιοποίηση και ε, λόγω και καταστάσεων σε γειτονικέ χώρε. Όλα αυτά απαιτούν ε, τέτοιε διαπραγματεύσει για την κατάρτιση αυτού του προπολογισμού και πραγματικά θέλω να συγχαρώ του συνεισηγητέ ε, που βρήκαν μία νέα προσέγγιση για το πώ μπορεί κανεί να πάει στι διαπραγματεύσει. Δηλαδή με σαφή προσφορά με σαφή μηνύματα. Δεν το είχαμε κάνει ακριβώς και δεν το είχαμε καταλάβει ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και για την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο αυτών των δείγματων. Πραγματικά λοιπόν συγχαρητήρια. Ταυτόχρονα ισχύει και το εξή. Ορισμένα τμήματα του προϋπολογισμού δεν έχουν τύχει της τέλειας διαχείρισης ε, και μιλάω και για τα κράτη-μέλη. Ε, που το βλέπουμε και στη συζήτηση. Ε, τι πόροι χρειάζεται να ε, εισαχθούν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το θέμα είναι η ανάγκη και δεν θα πρέπει να ξέρουμε τις πληγές. Θα πρέπει να δούμε αν πρέπει σίγουρα ε, να θεωρήσουμε υπεύθυνο και τον περιορισμό των εθνικών προπολογισμών, αλλά και το κατά πόσον τελικά έχουμε εκμεταλλευτεί και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αξιοποιήσει τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, φερθούν συγκεκριμένα κυρίω κράτη-μέρη με μεγαλύτερη συνέπεια και υπευθυνότητα. θέλουμε να μιλάμε για τέτοια πράγματα και για τα μεγάλα ταμεία, ε, για την αγροτική ανάπτυξη, για την συνοχή. Πολλά κράτη-μέλη, και μιλάω και για το δικό μου ομοσπονδιακό κρατήριο, ε, είχαμε μια, ένα, μια μεγάλη πρικοδότηση από την, ε, το Ταμείο Συνοχής και άμεσες πληρωμές προς την 2014 2014-2020. Αν χαθούν αυτά, Ουσιαστικά οι μισές επενδύσεις γίνανε από ευρωπαϊκά κονδύλια. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τα κλασικά κράτη συνοχής, αλλά μιλάμε και για άλλες ε, περιφέρειες σε μεγάλα κράτη. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν αυτό με τη συνοχή και είχα κάνει σε εκλογική περιφέρεια κάποια εργαστήρια, κάποια workshop ε, που μου έδωσαν ε, πάρα πολλά ε, στοιχεία για την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, τη τα κτλ. Και θα πρέπει λοιπόν να δράξουμε, να δράξουμε την ευκαιρία της, που μας έδωσε η Κομισιόν. Σίγουρα έχουμε το Brexit δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι ο λογαριασμός ε, της αποχώρησης. Εγώ τον βλέπω λίγο πιο ακριβό ε, από αυτό που βλέπουμε. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τις νέες ε, συμφωνίες. Αν δεν υπάρχει καθάριση μέχρι στιγμής των χρηματικών υποχρεώσεων δεν θα είναι αξιόπιστος ε, ούτε ε, έμπιστος ε, ο συνομιλητής μας εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο και μιλώ για τους φίλους Βρετανούς και το έχω πει και το ξαναλέω με απόλυτη ειλικρινία. Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και γι' αυτό σε αυτά τα μεγάλα ταμεία θα πρέπει να δούμε αν μιλάμε για ίδια ευθύνη, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ε, ειδικέ τάσεις αναχώρα, το βασικό κομμάτι, όχι τις ε, τεράστιες αυτές ε, εκθέσεις, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Και επίσης έχουμε και το κράτος δικαίου, που είναι και αυτό ένα θέμα που συζητούμε. Αλλά εκεί όλοι θα κρυθούμε. Ε, κανένας δεν μπορεί να φύγει ε, αυρόχης ποσή. Και θα ήθελα να δούμε και την απόφαση, την ετοιμιγορία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, μετά από μια καταγγελία του Φεβρουαρίου από Πορτογάλους δικαστές που είχαν ε, καταγγείλει τις περικοπές ε, στους μισθούς της και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έκανε δεκτή τα καταγγελόντες ότι στις δημόσιες υπηρεσίες σε καιρό κρίσης πρέπει να υποστούν περικοπές. Δεν έχουν οι δικαστές κάποια, δεν ανήκουν σε κάποια διαφορετική κατηγορία. Το πιο σημαντικό για μας βέβαια είναι τα συνοδευτικά σχόλια της απόφασης αυτής του δικαστή. Εγώ δεν είμαι νομικός, ε, έχω διαβάσει έτσι κάπως ε, στο περιθώριο γεωργικό δίκαιο, αλλά εδώ ε, διαβάσαμε πολύ ξεκάθαρα τι λέει και ο χάρτης για την Ευρωπαϊκή Θεγένεια, τους Ευρωπαίους πολίτες ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ανεξαρτησία των δικαστών. Αυτό λέγεται ξεκάθαρα. Ο χάρτης της Ένωσης είναι μέλος, ε, μέρος των συνθήκων, άρα ανήκει στο δίκαιο το ευρωπαϊκό και αυτό θα πρέπει να το δούμε και να δούμε και τι γίνεται ε, με τα κράτη-μέλη και συγκεκριμένα κράτη-μέλη δεν μπορούμε να παρακάμψουμε εμεί ε, στην Επιτροπή Προπολογισμών αυτά τα θέματα για το ποια είναι η διάθεση και η προδιάθεση των δημοκρατών απέναντι στο κράτο δικαίου. Ελπίζω μπορούμε να κινούμαστε και στο μέλλον μέσα στα, στο πλαίσιο αυτό των κοινωνικών. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε το 1,1 ε, κάτι ή το 1,3% και σίγουρα είναι λεπτό το θέμα ακόμη για πολλά κρατημέλη και κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει ε, να συνδέσουμε και κάτι που ίσως ε, δεν το έχουμε ακόμη επεξεργαστεί επαρκώς γιατί δεν έχει εκδηλωθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα κράτη-μέλη. Όταν δημιουργούμε έναν οργανισμό τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδεδρόμου. Για να σα φέρω ένα παράδειγμα. Τι επιπτώσεις, τι συμπεράσματα συνάγουν τα κράτη Γίνεται κάτι διαφορετικό. Αλλάζει η διοίκηση εθνική. Όχι, δεν αλλάζει. Έχουμε λοιπόν ε, ένα νέο ευρωπαϊκό οργανισμό, αλλά παραμένουν οι εθνικές δομές, άρα έχουμε επικάλυψη, έχουμε διπλά ε, όργανα. Ε, και τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Δεν συνάγονται οι επιπτώσεις και τα συμπεράσματα από τον τρόπο λειτουργία και τι αποφάσει των ευρωπαϊκών οργανισμών. Αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε και μαζί με το Συμβούλιο και μαζί με τα κράτη-μέλη και τα κοινοβούλια τεχνικά πρέπει να συζητήσουμε αυτό το πρόβλημα των διπλών-τριπλών δομών. Να δούμε μήπως κάπου έχουμε, το έχουμε παρακάνει και μπορούμε να ε, γυρίσουμε λίγο προς τα πίσω. Δεν είμαι υπέρ όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ούτε όμως λέω βέβαια ότι πρέπει και να κλείσουν όλα. Έρευνα. Ε, είχαμε μια ακρόαση για το θέμα. Είπαμε ότι έχουμε ε, πάρα πολλά προγράμματα, πάρα πολύ α, καλά, άριστα προγράμματα ερευνητικά που θα μπορούσαμε να τα τριπλάσια από αυτά που χρηματοδοτούμε τώρα να χρηματοδοτήσουμε, αλλά δεν έχουμε τους πόρους να το κάνουμε αυτό. Ίσως ε, πάλι ελλείψη ε, μέσων και πόρων στον εθνικό προπολογισμό να έχουμε ε, ανάγκη από αυτή την αύξηση του προϋπολογισμού για την έρευνα, κυρίως για την ανάπτυξη και μπορεί ίσως να πρέπει να ε, δώσουμε περισσότερα χρήματα και σε ό,τι αφορά ε, την προσέγγιση από τη μία έχουμε τη μετανάστευση και την ασφάλεια και από την άλλη έχουμε τη συνοχή. Δεν πρέπει να τα φέρουμε το ένα απέναντι στο άλλο. Έχουμε και τις, ε, το άρθρο 78 και 80. Τι γίνεται με την περίπτωση ενός μαζικού ρεύματος μετανάστευσης αλλά έχουμε ε, και ε, την ε, δίκαιη κατανομή. Το λέει το 80 αυτό. Μιλάει για ισομερή κατανομή και κάποιοι κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα. Το λέει όμως η συνθήκη, ξεκάθαρα. Επομένως, πράγματι, και με βάση αυτό το θέμα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την άποψη της Κομισιόν. Υπάρχουν χώρες που κάνουν περισσότερα. Ίσως και αυτά τα κράτη θα πρέπει να πάρουν λίγο περισσότερα κονδύλια, γιατί είναι και θέμα αξιοπιστία. Αλλά όχι ο ένας να στρέφεται εναντίον του άλλου. Ούτε να στρέφουμε τον ένα τομέα συνοχή απέναντι ε, αντίθετο με τον άλλον, παίρνοντα χάρη την άμυνα ή την ε, ε, μετανάστευση. Υπάρχει προσθέμενη αξία Έχουμε τις εθνικές δαπάνες που ουσιαστικά ε, δημιουργούν ένα ομοιόμορφο εντελώς ε, μοτίβο. Δεν ξέρω μήπως θα μπορούσαμε να μειώσουμε κάπως τις εθνικές δαπάνες όλες του κρατικό προπολογισμού. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες ε, διορθώσεις ώστε να αιτιολογήσουμε για να τεκμηριώσουμε αυτό που ζητάμε, το 1,3% και να μπορέσουμε να έχουμε ισοπέραση διαπραγματεύσει. Ah, Δεν κατάφερα να ανάψω το μικρόφωνο μου. Ευχαριστώ τον κύριο Μπέγκε για την έκκληση που μόλις απέκτηνε. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Γκαρδία Θαμπάλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές και δεν το κάνω τυπικά γιατί πραγματικά θεωρώ ότι έκανα εξαιρετική δουλειά. Κυρίως γιατί έδωσαν ουσία ε, στις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει τις μεγάλες πολιτικές και τις μικρές πολιτικές, αλλά οι συνεισηγητέ μας ε, ε, ξεκάθαρα δήλωσαν τι θέλουμε να πούμε όταν προσπιζόμαστε αυτές τις ε, πολιτικές. Για κάθε ένα από τα προγράμματα έχουμε ξεκάθαρη θέση και έχουμε να δώσουμε και ξεκάθαρη απάντηση σε όλες τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σεφής τρόπος εργασίας. Ιδίως γιατί δεν αφήνει περιθώρια για αυτοσχεδιασμούς και γιατί με τον τρόπο αυτό εργασία όλο το κοινοβούλιο, τόσο πάντων μεγάλη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, έχει μία θέση συνεπή και συντονισμένη. Η πρόταση των συνεισηγητών δείχνει και κάτι ακόμη. Δείχνει τη σοβαρότητα της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια σαφής πρόταση, αλλά είναι και τεκμηριωμένη, εμπεριστατωμένη το λέω ξανά, εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη. Αυτό θα πει bottom-up. Δηλαδή, πήγαμε και ξεκινήσαμε. Ποιε είναι οι ανάγκε. Τι προσθέσαμε τη μία με την άλλη. Και βάλαμε και ένα όριο. Και εργαστήκαμε με ένα σλόγγαν, αν θέλετε, με μία αρχή, ότι οι νέες προτεραιότητες ε, δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από περικοπές στι παραδοσιακές πολιτικές. Και αυτό ήταν, αυτή ήταν η του κύκλου, να φτάσουμε σε αυτό το 1,3 και γι' αυτό είναι και περιστατωμένε και τεκμηριωμένε προτάσει. Ε, γιατί θα μπορούσαμε να βάλουμε επιτάπητο στι ανάγκε αλλά τότε θα φτάναμε σε ένα προβλησμό 3, 4 και 5%. Γιατί η πολιτική συνοχή είναι όλο και πιο απαραίτητη και αν δούμε τις εκθέσεις περί ανισοτήτων θα δούμε ότι οι ανισότητες οξύνονται και δεν μειώνονται ούτε μεταξύ ατόμων ούτε μεταξύ ε, περιφερειών. Έχουμε και την έκθεση του ΕΕ για την κλιματική αλλαγή που μας έχει φέρει ενώπιον ε, τελεσιγράφου και θα πρέπει να δούμε και ποιο είναι το κονδύλι, δεν το έχουν προστοκοπήσει ακόμα, που θα πρέπει να διατεθεί για την αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή. Δεν είναι επαρκή, είμαι σίγουρη, σε σχέση με αυτό το οποίο προβλέπετε. Και υπάρχουν και άλλα θέματα που δεν ε, έχουμε ακόμα εκπληρώσει ε, απόλυτα του στόχου μα, άρα το 1,3 έχει νόημα. Θέλουμε να είμαστε και ρεαλιστέ. Γι' αυτό μείναμε σε αυτό το 1,3 που σίγουρα και δεν αρκεί. Και όταν μιλάμε για το δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και σε όλες τις γνωμοδοτήσεις εμείς ε, τονίσαμε σοσιαλιστές τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Στρατηγική και στόχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περί αυτού πρόκειται. Άρα θα πρέπει η βάση μας πάντα και γνώμονα με το βάση τον οποίο θα κινούμαστε θα πρέπει ακριβώς να είναι αυτή η στρατηγική. 1,3 100% βασίζεται, όπω είπα, στο ότι δεν θα περικοπούν προγράμματα για να χρηματοδοτηθούν άλλα. Πρόταση του Κοινοβουλίου ακριβώ είναι για να μην χρειαστούν περικοπέ, θα χρειαστεί αύξηση των ιδίων πόρων. Σε ό,τι αφορά τώρα του ίδιου πόρου, η πρόταση του Κοινοβουλίου νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα έχουμε καταθέσει ως γραπτή πρόταση, αλλά μπορεί να ε, χρειαστεί να είμαστε πιο συγκεκριμένοι χωρίς να επανεφεύρουμε κάτι καινούργιο σε σχέση με την έκθεση του Μαρτίου. Κάνοντας ένα βήμα πιο πέρα, με πιο συγκεκριμένα νούμερα, με πιο συγκεκριμένες προτάσεις, νομίζω ότι στο τμήμα των ιδίων πόρων μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την πρότασή μας, αλλά χωρίς σε καμία περίπτωση να αλλάξουμε τα ήδη συμφωνηθέντα. Σίγουρα μένει δουλειά στο μέλλον να γίνει, αλλά όπως είπα οι συνεισυχτές εργάστηκαν ε, με ιδιαίτερη αεφή τρόπο, καταθέτοντας έτσι αυτή την πρόταση με τόσο συγκεκριμένες προτάσεις και με πάρα πολύ καλά δομημένη απάντηση ε, στις προτάσεις Κομισιόν. Και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε και πιο εύκολο έργο στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κυρία Γκαρδία Σαμπάλ. Κανείς άλλος δεν ζητά το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στον εισηγητή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και μετά στον εισηγητή της Επιτροπής των Περιφερειών, οι οποίοι έχουν κληθεί να γνωμοδοτήσουν. Σε πέντε λεπτά θα είστε σε θέση να μας ε, μιλήσετε. Ναι, θα μιλήσω ισπανικά. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση που μας απευθύνεται να σας παρουσιάσουμε τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια της Επιτροπής μας στις 19 Σεπτεμβρίου. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η σημερινή σας συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουμε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους κυρίους Λεβαντόφσκι, Όλμπριχτ Ντεπρέ και την κυρία Τόμας, τους εισηγητές, γιατί έχουν διευκολύνει τη συνεργασία, ε, τις συναντήσεις για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε και εμείς τη γνωμοδότησή μας. Και θέλω να τους συγχαρώ επίσης για το εξαιρετικό κείμενο που μας παρουσιάζουν εδώ και που σας παρουσιάζουν, που είναι εναλλακτικό ε, κείμενο και έχει πολύ συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και συνάδει με τη βασική γραμμή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, όπου εμείς εγκρίναμε σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία και στο τμήμα των εργαζομένων και στο τμήμα των εργοδοτών και στο κοινωνικό τμήμα όλοι με τεράστια πλειοψηφία ε, τρέφουμε αυτή την ελπίδα να επηρεάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που κομίζουμε εδώ, δηλαδή έτσι ώστε να δώσει η Επιτροπή τους βασικούς πόρους για να υλοποιηθούν οι βασικές πολιτικές σήμερα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική συγκυρία την οποία διανύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στη γνωμοδότησή μας αναφέρουμε τους παράγοντες που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του για να δικαιούται να απαιτεί ένα προϋπολογισμό πολύ πιο φιλόδοξο και να υπάρχει αυτό το 1,3 του ΑΕΠ, του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Από το τέλος της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής και από την επόμενη χρονιά μέχρι το συνεχές έλλειμμα επενδύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους κινδύνους ε, του ε, εμπορικού προστατευτισμού που ε, βλέπουμε να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο μέχρι και τις τελευταίες εξελίξεις. Παντού λοιπόν βλέπουμε ότι συνεχίζεται η κοινωνική διάβρωση που είναι απότοκος της κρίσης και του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικοί διαχειρίστηκαν αυτή την κρίση. Και αυτό είναι και το πολιτικό στοιχείο το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το οποίο μας οδήγησε σε πολιτική κρίση και η εκδήλωση της πολιτικής κρίσης φαίνεται από την άνοδο των εθνικισμών της ακροδεξιάς το γεγονότος ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν πληρούν τις αρχές του κράτους δικαίου και μάλιστα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις γειτονικές μας χώρες και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια απάντηση με συνοχή και συνέπεια. Θέλει να υλοποιήσει αυτές τις πολύ διαφορετικές πολιτικές. Πρέπει να το δείξει αυτό και πρέπει να υπάρχει μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής ε, ε, Ένωσης ε, με μεγάλη φιλοδοξία, σε βάθος χρόνου, με μεγάλο εύρος, ή δελειώς θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι ανάγκη να υπάρχει συνέπεια και συνοχή με τις προτάσεις που διατυπώνονται εδώ. Πρέπει τουλάχιστον τα επίπεδα να διατηρηθούν, τα υφιστάμενα επίπεδα του υφιστάμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, να διατηρηθούν οι πόροι που απευθύνονται, που προορίζονται για τη συνοχή και τη γεωργική, τη γεωργική πολιτική. Και πρέπει να ενισχύσουμε ορισμένα κεφάλαια με τον προπολογισμό μας. Πρώτον, το τεράστιο κεφάλαιο των επενδύσεων και δεν μιλούμε μόνο για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αλλά όλα τα υποκεφάλαια και τα κεφάλαια του των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο προπολογισμό. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ειδικό πυλώνα, ειδικό κεφάλαιο για το πυλώνα των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να εκπληρώσουν τα κράτη-μέλη τους στόχους της ε, διακήρυξης του Γκέτεμπορκ, έτσι όπως υιοθετήθηκε αυτή πέρσι. Είναι απαραίτητο εντός μια στρατηγικής που θα διαμορφωθεί σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εντός αυτής της πολιτικής να διακρίνουμε συγκεκριμένες δράσεις έτσι ώστε να επιδιώξουμε και να πετύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τους στόχους της διακήρυξης του Γκέντεμπορκ για τα κοινωνικά εργασιακά δικαιώματα. Συμφωνούμε και θεωρούμε ότι για να έχουμε ίδιους σπόρους πρέπει να αναπτύξουμε όλες τις προτάσεις που ε, παρουσίαζε η ομάδα υψηλό επίπεδο υπό την ε, καθοδήγηση του Μάριο Μόντι. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση και σαφέστατα θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Η πρόταση είναι ανεπαρκής από πλευράς αριθμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και απορριπταία. Είναι θετική πρόταση με τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί, χρειάζεται όμως αύξηση και ολοκληρώνω εκφράζοντας τη συμφωνία μας με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Ο Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νικολά Τομπρόσλαβιτς για την Επιτροπή των Περιφερειών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μας δίνετε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών. Γνωμοδότηση που συντάξαμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ευκαιρία. Θα ήθελα συντομία να τονίσω ε, δύο-τρία στοιχεία της γνωμοδότησής μας. Η Επιτροπή των Περιφερειών αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυσκολεύθηκε, είχε μη δύσκολο καθήκον ε, κατά τη σύνταξη της ε, ε, σχετικής πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη διαφόρων θεμάτων και ιδιαιτέρως του Brexit. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή πλατφόρμα για βάση και βατήρας, εφαλτήριο για συζητήσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να συνεχιστούν πριν την οριστική έγκρισή της. Στηρίζουμε με τις επιλογές που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτεραιότητες, για τις προκλήσεις. Στηρίζουμε το αίτημα για την κατανομή και τη χορήγηση περισσότερων πόρων προς αυτό το σκοπό. Όχι όμως σε βάρος της συνοχής και της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Καλωσορίζουμε την πρόταση σύμφωνα με την οποία η χρήση των κεφαλαίων θα συνδέεται με την εφαρμογή του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη. Ζητούμε όμως να υπάρχουν σαφή κριτήρια για το, και κοινά κριτήρια για το πώς θα αξιολογηθούν αυτές οι ανεπάρκειες και οι τελικοί δικαιούχοι θα πρέπει να προστατεύονται εάν παρελπίδα και τελικά επιβληθούν κυρώσει σε ένα κράτος μέλος διότι η κρατική εξουσία δεν εφαρμόζει το κράτος δικαίου. Να μην είναι αυτό σε του τελικού δικαιούχου. Ε, Δεν θέλουμε ε, να είναι χειρότερη η θέση του τελικού δικαιούχου στο CPR, στη τελική απορρόφηση των κονδυλίων. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις περικοπές για την κοινή γεωργική πολιτική και ειδικότερα για το δεύτερο πυλώνα, ε, την ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαν απευθύνει έκκληση για υψηλότερους ίδιους πόρους. Αυτό θα έλυνε και το αίτημα να καλυφθούν νέες προτεραιότητες και νέες προκλήσεις από τη μία και θα διατηρούσε από την άλλη το μέγεθος της πολιτικής συνοχής και της κοινή γεωργικής πολιτικής στα υφιστάμενα επίπεδα το οποίο εμείς επιθυμούμε και το οποίο είναι το ελάχιστο που μπορούν να αποδεχθούν ε, οι οργανισμοί τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον κύριο εισηγητή από την Επιτροπή των Περιφερειών για τη σαφήνεια, τη συνέπεια ε, και την ε, ξεκάθαρη τοποθέτησή του. Πριν δώσω το λόγο στους συνεισηγητές, θα ήθελα για άλλη μια φορά να εκφράσω το θαυμασμό που τρέφω προς τα πρόσωπά τους και να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς αυτούς. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σβάρτς, λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε ένα έγγραφο που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεκινήσει στις βέλτιστες δυνατέ συνθήκε και προποθέσει τη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Ελπίζοντα ότι αυτό το Συμβούλιο θα καταφέρει να καθορίσει μια εντολή διαπραγματευτική πριν το τέλο του 2018. Επιτρέψτε μου να επιμείνω στην έννοια τη Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και στην έννοια των προκλήσεων που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση και στι οποίε θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε επίπεδο κλιματική αλλαγή, άμυνας, ασφάλειας, ψηφιακής οικονομίας, μετανάστευσης, πολιτικής για το διάστημα, μεταξύ άλλων. Όπως ε, το είπε και ο κύριος Μπέγκε, για τις διάφορες υπηρεσίες ε, που έχουμε συγκροτήσει και συστήσει, Συχνά βλέπουμε ότι κάποιες δαπάνες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο δεν έχουν πλέον καμία αποτελεσματικότητα και θα ήταν αποτελεσματικές αν γίνονταν ως μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού σχεδίου. Άρα πρέπει να απευθύνουμε μια έκκληση, ένα κάλεσμα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για να έρθουν σε συμφωνία, για να θεσπίσουμε και να θεσμοθετήσουμε αυτό το οποίο αποκαλούμε ευρωπαϊκό κοινό αγαθό και το οποίο πρέπει και μπορούμε να υπερασπιστούμε προς όφελος και προς το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη, κάτι το οποίο θα δείξει την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Εάν ταυτίσουμε και αναγνωρίσουμε τις δαπάνες οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές όταν γίνονται σε εθνικό επίπεδο γιατί οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, τότε εύκολα διανοείται κανείς ότι αυτές οι δαπάνες θα φύγουν από το εθνικό προϋπολογισμό, δεν θα τον βαραίνουν, θα βαραίνουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα γίνει ακόμα πιο στεναρό, χωρί όμω να αυξήσουμε τη δημόσια δαπάνη στην Ευρώπη και έτσι θα δείξουμε ποια είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αφού θα είναι δαπάνες που θα αναλυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να βαρύνουν περαιτέρω τον ε, εθνικό φορολογούμενο του κάθε κράτους μέλους. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σβάρτς. Θέλω να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία του σχεδίου έκθεση, την διάμεση. Αυτή. Θεωρούμε ότι είναι καλή βάση για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αυτήν η διάμεση έκθεση και θέλουμε να συγχαρούμε τους τέσσερις εισηγητές. Βέβαια, το τελικό ποσό είναι φιλόδοξο, 1,3% του καθάριστου του εθνικού εισοδήματος. Καλό είναι αυτό βέβαια, ότι υπάρχει φιλοδοξία. Και αυτός είναι και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άλλωστε. Έχετε αυξήσει την αξιοπιστία της έκθεσης κάνοντας αυτή την πολύ αναλυτική κατανομή για το πώς ε, θέλετε το 1,3% να οδηγήσει για ορισμένα προγράμματα. Και νομίζω ότι και αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα τη συζήτηση που ήδη έχει ξεκινήσει το Συμβούλιο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει και αυτά που λέτε για αρκετά οριζόντια ζητήματα. Δεν θα τα καλύψω όλα. Ε, επιλέγω ένα σημαντικό, που είναι η ευελιξία. Η έκθεσή σας βασίζεται στην πρόταση της Κομισιόν για ευελιξία και ζητάτε μεγαλύτερη ευελιξία, κάτι το οποίο είναι κατανοητό. Δυστυχώς όμως στο Συμβούλιο η συζήτηση πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη, ομάδες κρατών ε, μελών που θέλουν ε, την ευελιξία, το μέσο ευελιξία, ε, να συγχωνεύσουν πολλά από αυτά τα μέσα. Και αυτό σίγουρα θα μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ευελιξία. Και νομίζω ότι ξέρουμε πολύ καλά τι έδωσε στο PDP η ε, πρόταση που διαπραγματεύτηκε το Κοινοβούλιο κυρίως ε, με το μέσο ευελιξίας ε, που βοήθησε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τη μετανάστευση και και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό και να το θέσετε στις ε, συνομιλίες σας με το Συμβούλιο. Για τους ίδιους πόρους επίσης ε, ευπρόσδεκτα αυτά που λέτε και τα μηνύματα τα λάβαμε ξεκάθαρα και αυτό το σύνδεσμο που κάνετε με το πουδουπού και το μερίδιο των ίδιων πόρων και αντιλαμβανόμαστε πλήρως ε, την αρισιμότητα όπως συνέθεσε ο κύριος Λεβαντόφσκι. Σημειώνουμε επίσης, ο Επίτροπος Έτιγκερ το έχει πει επανειλημμένος σημειώνουμε άλλους πιθανούς υποψηφίους ε, όπως το FTT ή το ψηφιακό φόρο για υποψήφιους ως ίδιους πόρους ενώ νέους φόρους. Θα συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, έχουμε προχωρήσει το έργο μας για βασικές πράξεις ό,τι αφορά αυτούς τους δύο φόρους, τον ψηφιακό και το FTT φόρο ψηφιακών συναλλαγών. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που υποστηρίζετε το μηχανισμό κράτους δικαίου. Θα ήθελα όμως εδώ να κάνω μια διευκρίνηση επειδή συζητήθηκε και το έθεσε κυρίως το θέμα η κυρία Γκρέσλε. Το άρθρο 4.2 του σχεδίου κανονισμού προτείνουμε πράγματι προστατεύει τους τελικούς δικαιούχους. Άρα συμφωνούμε με σας και την ανησυχία σας και το λέμε στον κανονισμό. θα μπορούσαμε ίσως να σας καλέσουμε να σκεφτείτε κατά πόσον εσείς αυτό θέλετε να το λέτε μηχανισμό επιβολής κυρώσεων. Η νομική βάση όπως γνωρίζετε για το μηχανισμό κράτους δικαίου είναι η, γης, είναι η χρηστή συγγνώμη, διαχείριση. Δεν το θεωρούμε κύρωση αυτό. Ε, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για μα είναι ένα προφανή, αυτονόητο τρόπο διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο μια συνδιαχείριση και ένα μηχανισμό επιβολή κυρώσεων υπό την έννοια αυτή γίνεται ιδιαίτερα σκληρό ω διατύπωση όταν μιλάμε για διαχείριση του υπολογισμού κατ' ουσίαν. Πράττω με τι ευκαιρίε για να σα ενημερώσω ε, για τη διαδικασία, πώς θα συνεχιστεί. Έχουμε στο Κόρεπερ συνάντηση αυτή την εβδομάδα για κάποια οριζόντες δήματα μεταξύ των οποίων και ευελιξία, όπως προείπα, κατηγορία 13-5-7. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και γεύμα εργασίας, ε, γεύμα εργασίας για τα θέματα αυτά και το debriefing του Κοινοβουλίου ε, όπως προβλέπετε θα επακολουθήσει. Γρήγορα προχωράμε στο Συμβουλίο, σε τεχνικό επίπεδο, δύο συναντήσεις την εβδομάδα και εξέταση των ζητημάτων. Και φυσικά η έκθεσή σας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον Νοέμβριο, οπότε το Συμβούλιο και η Κομισιόν βέβαια θα ενημερωθεί για τις θέσεις. Ολοκληρώνω εδώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπουμε στις επόμενες συζητήσει για την έκθεση. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur Schwartz. Merci d'avoir souligné l'ambition du Parlement. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σφάρτς, που τονίσατε και την ε, φιλοδοξία από πλευράς ε, κοινοβουλίου. Δεν δείχνει την ευελιξία, βέβαια, το Συμβούλιο. Τώρα έχουμε τις νομικές βάσεις που έχουμε. Από πολιτικής πλευράς όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι φορολογούμενοι ορισμένων κρατών που είναι καθαροί εισφορείς θα εκπλαγούν αν δουν ότι δεν σέβονται τον Ευρωπαϊκό Χάρτη ε, αυτά τα κράτη. Και αυτό θα βαρύνει και στι προσεχεί ευρωεκλογέ κατά πάσα πιθανότητα. Δεν υπάρχουν μόνο λοιπόν οι νομικέ πτυχέ. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Ευρώπη είναι ένα οικοδόμημα που εδράζεται σε κοινέ αξίε, σε ελευθερίε και στο κράτο δικαίου. Κύριε Μπέγκε, θέλετε το λόγο. Νομίζω τελικά, κύριε Πρόεδρε, προτάσει που συζητήσαμε σήμερα δεν είναι μόνο φιλόδοξε, αλλά είναι και λογικέ. Και νομίζω ότι η Κομισιόν αυτό θα πρέπει να διατηρήσει, να συγκρατήσει τη λέξη λογικέ προτάσει, όχι φιλόδοξες προτάσεις. Ωραία, λοιπόν, απευθύναμε και αυτήν την ε, έκκληση προ την ε, Επιτροπή. Μην ακούσει τα κράτη-μέλη που δεν θέλουν να πληρώσουν τίποτα. Το θέλουμε είναι τι θέλουμε να κάνουμε. Να δώσουμε μια, την εικόνα μια ευρώπη αδυναμη ή μιας Ευρώπης που μπορεί να είναι κυρίαρχη και αυτόνομη, που στρατηγικά να είναι ανεξάρτητη. Εάν δεν το προσφέρουμε αυτό στους Ευρωπαίους πολίτες, πώς να τους πούμε ότι θέλουμε μια Ευρώπη που θα προετοιμάσει το μέλλον μας και θα μας προστατεύει. Κυρία Τομα, κύριε Όλμπριχτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και την Επιτροπή των ε, Περιφερειών και την ΕΟΚΕ, όχι μόνο για τις γνωδήσεις τους, αλλά για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Σας ευχαριστούμε. Είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολλά τα σημεία σύγκλησης μεταξύ μας. Προτού δώσω το λόγο στον κύριο Όλμπριχτ για τα πρώτα συμπεράσματα, να πω ότι τόσο πολύ ήθελα να εξεργήσω καλά την μεθοδολογία μας που ήθελα να κάνω σχόλια περί της πολιτικής μας. Το πράγμα που θα κάνω τώρα. Ε, κρίμα που μερικοί από τους συναδέλφους που εξέφρασαν απορίες έφυγαν εντωμεταξύ. Για τους ε, ε οριζόντιους στόχους ε, δεν ε, μείναμε, δεν περάσαμε σε λεπτομέρειες, αλλά παραμείναμε στις προτεραιότητες του 30% όπως εκπαιδευόταν στην ε, απόφαση του Μαρτίου. Ακολουθήσαμε αυτή την αγκάρσια προσέγγιση γιατί στην έκθεση της συναπόφασης προβλεπόταν σε μια τροπολογία στην ενδιάμεση αναθεώρηση που αυτή τη φορά είναι υποχρεωτικό να γίνει, κάτι που θα μας γλιτώσει από συζητήσεις για το αν είναι υποχρεωτική ή όχι, πώς θα πρέπει να δούμε τα πράγματα και πότε, θα είναι υποχρεωτική, οπότε να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε, γιατί θα πρέπει να έχετε κάποιο πίνακα αναφορά όχι αφηρημένων επιδόσεων, αλλά συγκεκριμένων επιδόσεων που να λαμβάνουν υπόψη του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπω και τη ισότητα ε, ανδρών γυναικών. Που σωστά μα ε, εξέθεσε η νεαρή κοπέλα που έφερε εδώ ο κ. Τόρβαλτ και μα σύστησε η ισότητα ανδρών και γυναικών, α πούμε, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Ή για τα θέματα τη ευελιξία. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει να βρούμε την μέση οδό μεταξύ ευελιξία και τη προβλεψιμότητα και των πολιτικών στόχων, διότι θα μπορούσαμε να έχουμε έναν απολύτω ευέλικτο προπολογισμό, αλλά τι θα ήταν αυτό, χωρί πολιτικού στόχου και χωρί πολιτικέ προτεραιότητε. Αλλά θα μπορούσε να προσαρμόζεται σε ό,τι συμβεί σε ό,τι μας αρέσει και σε ό,τι προκύψει ω προτεραιότητα ανά πάσα στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν και ευελιξία και προβλεψιμότητα αλλά και πολιτική στόχη. Και έπειτα θα συνεχίσω να προσπαθώ να πείσω τον κύριο Κέλμελ και θα προσπαθώ στο τέλος της θητεία. Θα προσπαθώ να σας πείσω ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς στα επιχειρήματά μας. Και για να υποστηρίξω τα επιχειρήματά μου, θα σας, δώσω την, ε, ε, θα σας αναφέρω την έκθεση της ε, Βουλής, της Ομοσπονδιακής Βουλής. Είναι σαφής. Λέει ότι πρέπει να μην γίνουν περικοπές στην πολιτική συνοχή, ότι δεν πρέπει να γίνουν περικοπές στην πολιτική γεωργία, ιδίω στο δεύτερο πυλώνα. Τι να πω, εντάχει διαβάζοντα την έκθεση της Bundesrat, έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για έκθεση που αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, ούτε τόσο πολύ διαφωνούμε. Μάλλον θα τα καταφέρουμε. Και τέλος, για τα προγράμματα τα ίδια που είναι και ουσία. Με συγχωρείτε. Ε. Τα λέτε μετά μεταξύ σας για τα προγράμματα και την πρικοδότησή τους. Να θυμίσω στην κυρία Γκρέσλε ότι προφανώς δεν είμαστε εμείς ε, οι εμπνευστέ και αυτοί που ε, κάνουμε να λειτουργούν τα περισσότερα προγράμματα. Μάλιστα τα αναθέσαμε στις επιμέρους ε, επιτροπές, όπως έγινε με το Child Guarantee, την εγγύηση για τα παιδιά. Αλλά για αυτό το νέο πρόγραμμα, ας πούμε, μου φαίνεται σαφές τι συμβαίνει από πού προέρχεται, ε, οφείλεται στο γεγονό ότι από την ε, υλοποίηση, των, ε, την εφαρμογή πολιτικών λιτότητα στην Ευρώπη και μετά, υπάρχει δραματική αύξηση τη φτώχεια, ιδίω στην ομάδα ηλικία των παιδιών και των υπείων. Είναι ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί σε πολλές χώρες και πρέπει να το ανακόψουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την παιδική φτώχεια και υποθέτω, δεν το υποθέτω απλώς, το γνωρίζω γιατί υπάρχουν πολιτικά πιλωτικά προγράμματα τα οποία έχει οργανώσει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Νομίζω μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο αυτών των πιλωτικών προγραμμάτων. Ως προς τους μηχανισμούς ε, διασύνδεση, κάποιο έθεσε την ερώτηση, νομίζω, ε, εδώ προβλέψαμε αύξηση 6 δις Βεβαίω ε, είναι περιορισμένο το χαρτοφυλάκιο, αλλά είναι ένα βήμα πρόοδου. Και για να ολοκληρώσω για την πολιτική μας και σε σχέση με όσα είπε και ο κύριος Φερνάντε, Ιδίω για το Συμβούλιο. Όπως είπατε και εσείς κύριε Φερνάντε και άλλοι, δουλειά, ε, σκοπός του Κοινοβουλίου είναι να κάνει τη δουλειά του στα δυνατόν καλύτερο και να αναλάβει τι ευθύνε του και τις πολιτικές του ευθύνε όμως ε, που απαιτούν από τη μια να έχουμε προπολογισμό στο ύψος των ε, προσδοκιών των πολιτικών που διαφημίζουμε για να σταματήσουμε αυτή την υποκρισία που έχει να κάνει με το να ανακοινώνουμε προτεραιότητες τις οποίες δεν χρηματοδοτούμε, μετά κάνουμε περικοπές. Ό,τι έχουμε τώρα στο τωρινό τα δημοσιονομικό πλαίσιο με την πολιτική της έρευνας ας πούμε. Τι έγινε, προσαρμόσαμε τα κονδύλια στις προτεραιότητες, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα κονδύλια στις προτεραιότητες που ε, ανακοινώνουμε. Και έπειτα, συμφωνώ, ε, η θέση μας είναι απλώς λογική. Είμαστε απλώς μετριοπαθείς και λογικοί και σοβαροί. Αυτό που δεν είναι σοβαρό και με συγχωρείτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το 1,8 1,08 ε, του, ε, του ΑΕΠ ε, θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν. Θυμηθείτε τι γινόταν την δεκαετία του 1990. Είμαστε στο 1,27%. Γιατί λέμε ότι το 1,3 είναι υπέρμετρο, φιλόδοξο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είχαμε την δεκαετία του 1990 τα προβλήματα τη κρίση που πρόκειται μετά το 2008. Δεν είχαμε τα προβλήματα τη ασφαλεία και τη άμυνα. Δεν είχαμε την ανεργία των νέων ιδίω. Δεν είχαμε πρόβλημα με τη φτώχεια των παιδιών που μόλι ανέφερα. Ε, δηλαδή με λίγα λόγια δεν είχαμε τόσες πιέσεις, απειλές ε, και κάτι που να μας υποχρεώνει να σοβαρευτούμε επιτέλους. Είχαμε άλλα challenge και είχαμε 1,27% του ΑΕΠ. Τώρα 1,08% ε, ε, τόσα χρόνια μετά είναι σοβαρό αυτό. Δεν είναι σοβαρό το 1,08%. Ε, αυτό που είναι σοβαρό είναι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι τελικά αυτή θα προκριθεί στα μέσα Νοεμβρίου, ε, τουλάχιστον αφού ψηφίσει και ολομέλεια. Με αυτά θα ολοκληρώσω, διότι πραγματικά, και το είπα και λίγο προηγουμένω, αλλά αυτό που πραγματικά με κάνει να θέλω να αντιδράσω είναι ότι στι διμερεί ε, συζητήσει με εκπροσώπου των κρατών μελών έχω την εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη και είπα, ε, είδα με την έκθεση του Ισμπούντες, αλλά και από τη Δημοκρατία της Τσεχίας, από το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, από την Πορτογαλική Βουλή. Άμα διαβάσω τις θέσεις τους, τις θέσεις των εθνικών συνελεύσεων ε, στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, πραγματικά μου δίνεται η εντύπωση ότι βρισκόμαστε ακριβώς στα όρια, στο μέτρο της λογικής, στο, στο στην μέση οδό, ακριβώς αυτό που είναι λογικότατο. Δηλαδή είναι σαν να γυρνάνε όλοι να μας πούνε ε, ναι, με το, με το κοινοβούλιο συμφωνώ, αλλά δεν βλέπω γιατί υπάρχει αυτή η αδράνεια μετά, αυτή η έλλειψη ανάληψης δράσης. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπερασπιστούμε με σοβαρό και εύστοχο τρόπο τις θέσεις μας και σε κάθε περίπτωση να συνεχίσουμε να πιέζουμε τα κρατή ένα προς ένα. Ε, επιτέλους, το είπα τις προάλλες, τον εκπρόσωπο και των κάτω χωρών. Πείτε τα στο Κοινοβούλιο. Βγείτε από τον κύκλο του Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν θα έρθει να το κάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει κάπου να ξεμπερδεύουμε με αυτές τις παλιές προκαταλήψεις που είναι εντελώ ξεπερασμένες των ε, χειρών και οδοφραγμάτων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Όχι, ας έχουμε πολιτικές συνδιαλλαγές μεταξύ των και των ΔΕ. Και ίσως και να καταφέρουμε μέχρι το τέλος της θητείας να έχουμε μια φιλόδοξη θέση και σοβαρή και αξιόπιστη και στο ύψος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Είναι θέμα διακυβέρνησης όλα αυτά. Είναι Είναι σαν την αρχίστρα. Μπορεί να είναι ατομικά οι μουσικοί πολύ, να παίζουν πολύ καλά το όργανο του ο καθένας, αλλά πρέπει να είναι συλλογικό ο ήχο για να είναι καλός. Ο κύριος Όλμπρεχτ παρακαλώ. Είναι αυτή η συζήτηση για τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά που λένε τα κράτη-μέλη ότι θέλουν να κάνουμε την κοινή πολιτική είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο, πόσο θα στοιχήσει και τρίτον, έχουμε τα χρήματα γι' αυτό. Όταν συζητούμε για ένα από αυτά τα χρόνια, ε, λέμε σαν κοινοβούλιο ότι πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε μαζί και λέμε ότι ε, το κόστος είναι τελικά το 1,3. Έτσι προκύπτει αυτό το 1,3. Και αυτή είναι η λογική πίσω από αυτό το σκεπτικό. Τα όρια από το 1,0 που θέλουν κάποια κράτη-μέλη και το 1,3 που θέλουμε εμείς υπάρχουν. Η Κομισιόν όμως δεν είναι στο μέσο μεταξύ 1,0 και 1,3. Η Κομισιόν τίνει προς το 1,08. Άρα δεν είναι εύκολη θέση στρατηγικά για τις διαπραγματεύσεις. Εμείς συμπεριφερόμαστε ε, φυσιολογικά. Ας είμαστε και ορθολογιστές. Ας σκεφτόμαστε με λογική και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν συζητά κανείς τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες και όταν διαβάζει ανάμεσα από τις γραμμές αντιλαμβάνεται ότι εμείς εκφράζουμε αυτά που λένε οι συνάδελφοι. Όταν ο κύριος Σολέ είπε ότι για μας το σημαντικό δεν είναι ποια μέρα θα κλείσει η συμφωνία πριν ή μετά τις ευρωεκλογέ, αλλά το περιεχόμενο αυτής συμφωνούμε όλοι. Και εμείς ε, ε, χρειαζόμαστε προϋπολογισμό με καλή ποιότητα. Δεν είναι ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου για μια μέρη, αλλά δεν θα το στείλει το, το Συμβούλιο για έγκριση εάν ξέρει ότι δεν θα το εγκρίνουμε. Εκτός και αν θέλει να προκαλέσει καταστροφή, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ο χρόνος απαιτεί την καλή ποιότητα. Ποια είναι η καλή χρονική συγκυρία σε πολιτικό επίπεδο. Ποια προσέγγιση απαιτείται. Όλα αυτά είναι τα βασικά. Και είναι επίση ενδιαφέρον το γεγονό ότι ορισμένοι συνάδελφοι από το EFTD για παράδειγμα λένε ότι κάποιε από τι εκτόσει πρέπει να παραμείνουν. Αυτό είναι καινούριο τώρα. Ποιε εκτόσει η Ολλανδική, η Γερμανική, κάποια νέα. Αυτά αλλάζουν τη φιλοσοφία μας τελείως, το πνεύμα. Ε, δείχνουν όλα αυτά πόσο δύσκολη θα είναι η συζήτηση και εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις και όσο πλησιάζουμε στι ευρωεκλογέ, τόσο θα οξύνονται οι διαφορές. Δύο είναι τα βασικά. Πρώτον, κράτο δικαίου. Βεβαίω, έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Γκρέσλε. Δεν είμαστε καθόλου αφελεί ως πολιτικοί όμως, ποιος θέλουμε να νιώσει τις συνέπειες. Οι κυβερνήσεις και να πληρώσουν από τον εθνικό προπολογισμό ή ο τελικός δικαιούχος, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Αυτές θα το νιώσουν. Θα το νιώσουν ότι κάτι πάει στραβά και είναι ο μόνος τρόπος να κάνουμε τις κυβερνήσεις να αλλάξουν. Ω πολιτικοί λέμε α μην υπερβάλλουμε, γιατί αν κάνουμε τον αντίκτυπο να το νιώσουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, τότε οι αντιευρωπαϊστές ε, θα βιώσουν τη χρυσή τους εποχή. Πρέπει να δούμε και τους πολιτικούς συσχετισμού. Όλοι θα είναι έξαλλοι. Άρα α είμαστε σαφέστατοι. ποιο παραβαίνει την νομοθεσία Ποιο δεν διορθώνει το σύστημα. Η απάντηση είναι οι κυβερνήσει. Άρα οι κυβερνήσει πρέπει να είναι υπεύθυνε και να φέρουν την ευθύνη. Ο, και υπόλογε. όχι έναντι τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έναντι των πολιτών τους, έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να τη νιώσουν την ευθύνη αυτή. Για αυτά που είπε ο, ο στο πάνελ, στα αριστερά του Πρόεδρου. Το SAFE δεν είναι στόχος, είναι ένα καλό εργαλείο. Είπατε ότι ένας από τους στόχους προτεραιότητας είναι το SAFE. Όμως δεν θα αντικαταστήσει τα πάντα. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα για να γίνει διασυνοριακή και εγκάρσια και ευρεία συνεργασία κτλ. Συμφωνώ. Όμως η συζήτηση μεταξύ της Επιτροπής Τραν και της Επιτροπής Ρέτζι για το ότι το Ταμείο Συνοχής θα μεταφερθεί στο ΣΕΦ πρέπει να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Αν πάρουμε χρήματα από την πολιτική συνοχή και τη βάλουμε στο safe και μείνει για τρία χρόνια στους εθνικούς φακέλους, αυτό είναι διαφορετικό. Εάν το πάρουμε από το safe και μπει σε ελεύθερο ανοιχτό διαγωνισμό τότε κάποια κράτη-μέλη θα ενδιαφερθούν για αυτό το σύστημα γιατί θα είναι έτοιμα και ξέρουν ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν θα ενδιαφερθούν γιατί δεν είναι έτοιμα, άρα θα τα πάρουν τα χρήματα και έτσι τα χρήματα θα φύγουν από τη μία χώρα και θα πάνε στην άλλη χώρα. Και δεν θα πω ποια χώρα το παλεύει να το πετύχει αυτό, αλλά την ξέρετε. Ορισμένε χώρε το περιμένουν αυτό. Να φύγουν τα χρήματα από το Ταμείο Συνοχή, να πάνε στον ανοιχτό διαγωνισμό και έτσι κάποιε χώρε θα πάρουν χρήματα που προορίζονταν για άλλε. Έτσι έχει η πραγματικότητα. Αυτό, γι' αυτό διαγωνίζονται. Και έχω και ένα ερώτημα προς τον κύριο Κόλμερ. Ξέρω τον τρόπο που σκέφτεστε. Συμφωνούμε στη διάγνωση, αλλά δεν συμφωνούμε στα συμπεράσματα. Καλώς. Αλλά ε, το ερώτημά μου είναι πολύ πολιτικό. Η ομάδα σας θα συμφωνήσει με τη μείωση των πόρων για το Ταμείο Συνοχής και τη Γεωργία. Εσείς τι παρασιά... Εγώ εκπροσωπώ την πλειοψηφία των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Και από το ΕΛΚ έχετε διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Όμως είναι πολύ ριζοσπαστική η προσέγγισή σας. Ε, έχουμε μικρέ διαφορές, αλλά είναι σημαντικό από πολιτικής απόψεως. Αυτό έχω να πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο τους, στους συνεισηγητές των ιδίων πόρων. Ο κύριος Λεβαντόφσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις με αρχική την πιο σύντομη. Στις 16 Οκτωβρίου, μετά το μεσημεριανό γεύμα, θα πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε μάθει περισσότερα για το κατά πόσο τα κράτη-μέλη κινούνται περισσότερο προς μια κοινή θέση ή συνεχίζουν να τοποθετούνται για να έχουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Ας ελπίσουμε ότι ε, τότε θα είναι το κλίμα πιο ευνοϊκό προς τη διαπραγμάτευση. Τώρα, για τους ίδιους πόρους, θα πρέπει συνεχώς να επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τις αρχές που κρύβονται πίσω από την πρότασή μας. Πλήρη σεβασμό στην φορολογική εθνική κυριαρχία των κρατών μελών πρέπει να είναι ομόφυλον η απόφαση που κυρώνεται από τα εθνικά κοινοβούλια και αν υπάρξουν κάποιοι ήδη πόροι, αυτό δεν είναι απότοκο στον συσχετισμό μεταξύ διαφορετικών ειδών φορολογίας για ε, διαφορετικό μέρος των εθνικών εσόδων από φορολογία που πάνε προς το κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά είναι κάποιες νέες υποψήφιες πηγές και η συνεισφορά GNI του Εθνικού Ακαθάριστου Εισοδήματος που θα πρέπει να παραμείνει, γιατί ήδη οι πόροι είναι απρόβλεπτοι, δεν μπορούν να προβλεφθούν, ενώ ε, ε, τα, οι εθνικοί προπολογισμοί είναι πολύ προβλέψιμοι και λειτουργούν σταθεροποιητικά. Εξού και υπάρχει η αιρεσιμότητά μας για τα έσοδα από δαπάνες και, ε, και τα, θα πρέπει εκεί η διατύπωση να είναι πολύ προσεκτική για να μην, για να μην πέσουμε σε παγίδα στη συνέχεια. Εάν τελικά ολοκληρωθεί και δημιουργηθεί και εφαρμοστεί το κακό σενάριο. Τώρα, να, έχουμε, να, να συμπληρώσουμε την μακροοικονομική ερεσιμότητα αιρεσιμότητα και τη διαδικασία βάσει του άρθρου 7, η οποία δεν είναι πολύ ισχυρή αυτή τη στιγμή. Όταν έχουμε εργαλειοθήκη κυρώσεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνουμε ότι θέλουμε να τιμωρήσουμε τους πολίτες και όχι τους ε, κυβερνήτες και τις κυβερνήσεις που έχουν παραβεί τους κανόνες. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα να αναπτύξουμε μια νέα μεθοδολογία διάσωσης των τελικών δικαιούχων. Εάν οι κυβερνήσεις πρέπει να πληρώσουν σε περίπτωση αναστολής των ευρωπαϊκών κονδυλίων ε, δεν τα βάζουν από την τσέπη τους, τα βάζουν από τα χρήματα του φορολογούμενου. Άρα περί ε, του ιδίου πρόκειται, περί των χρημάτων του φορολογούμενου πρόκειται. Αλλά ας προσπαθήσουμε να καταστήσουμε πιο ορατό ε, στον Ευρωπαίο πολίτη ότι δεν θα πρέπει να τιμωρείται ο ίδιος για την απροσεξία ή την απερισκεψία της κυβέρνησής του. πρόεδρος. της Δημοκρατίας μας η κυριαρχία είναι λαϊκή και οι κυβερνήσεις προέρχονται από την ψήφο των πολιτών. Άρα υπάρχει και ευθύνη του πολίτη που ψηφίζει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ περίπλοκο όλο αυτό. Να ε, και τιμωρήσει κανείς μια κυβέρνηση και να γλιτώσει από την τιμωρία τους ψηφοφόρους και τους πολίτες που την εξέλεξαν. Ο κύριος Σάρβαμα. Ευχαριστώ. Τελικά, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς 100% να διαχωρίσει την κυβέρνηση από το λαό που την εκλέγει, όσο την και είναι αυτό. Αυτό είναι και το βασικό αυτού του εγχειρήματος. Σας ευχαριστώ που εξεφράσατε με πιο εύγλωτα λόγια τις δικές μου σκέψεις, ο κύριος Ντεπρέ. Εν συντομία κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που μπόρεσαν να στηρίξουν τις προτάσεις μας. Σημειώνω ότι ορισμένοι εξ αυτών έχουν την πρόθεση να υποβάλουν ε, τροπολογίες τις οποίες θα εξετάσουμε με τη δέουσα προσοχή προσπαθώντας να πετύχουμε το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ αυτού που θα δείξει την αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του στοιχείου σοφροσύνης και προσοχής και επιμέλειας στις διαπραγματεύσεις για να μην βρεθούμε σε μια απριόρη κατάσταση αδιεξόδου. Επομένως η ισορροπία που θα πρέπει να βρούμε θα είναι απότοκο της λειτουργία ενό εξαιρετικά περίπλοκου μηχανισμού. Ω εισηγητής τη ομάδα μας και συνεισηγητής για τους ίδιους πόρους, οφείλω να πω ότι ε, διακατέχομαι από πλήρη αποφασιστικότητα και συμμερίζομαι πλήρως ε, τα λεγόμενα ορισμένων συνεδέλφων. Η συζήτηση όμως μόλις έχει ξεκινήσει. Εάν εδώ δεν έχουμε συμφωνία, το ίδιο θα συμβεί και σε επίπεδο κοινή γνώμη. Αυτό που αποφασίζουμε σήμερα είναι μια πολιτική απόφαση, μια πολιτική επιλογή και μια πολιτική μάχη, γιατί πρέπει να πείσουμε. Στη δική μου πολιτική ομάδα έχουμε βουλευτές που λένε ότι δεν ε, μου αρέσει το Brexit, αλλά θα γίνει. Δεν... Ε, ε υπάρχει ένα κράτος που απουσιάζει, άρα να πάρουμε ε, τις δαπάνες που προορίζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θέλετε να μας λένε Θέλετε να αναπαράγετε τις ε, πολιτικές χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τις εξελίξεις στο παγκόσμιο σκηνικό. Ε, θέλετε να προστατεύετε τη γεωργία για παράδειγμα και δεν βλέπετε τον ανταγωνισμό ε, και τις πιστώσεις που πρέπει να δοθούν για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή μετάβαση. Παντού σε όλες τις πολιτικές ομάδες υπάρχουν αυτοί οι παμπόνηροι. Έχουμε κάνει τις επιλογές μας, τι υιοθετώ και θα τι υπερασπιστώ. Όμως και εντός πολιτικών ομάδων η συζήτηση θα είναι ε, ένθερμη και δύσκολη και ζωντανή και αυτό είναι καλό ε, μήνυμα για τη δημοκρατία ε, και είναι ένα καλό μήνυμα έτσι ώστε πράγματι ο δημόσιος διάλογος με την εμπλοκή και τη συνεισφορή της κοινή γνώμης να διεξαχθεί και να αποκτήσει πολύ περισσότερη ορατότητα από ό,τι σήμερα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Πράγματι, Μακάρι να μπορέσουμε να έρθουμε σε συμφωνία μεταξύ μας και αυτό πρέπει να το δούμε σε επίπεδο κάθε πολιτικής ομάδας και όντως κάποιες πολιτικές ομάδες δεν είναι τόσο ομοιογενείς αλλά ετερογενείς στις διατυπώσεις τους. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό μέτωπο και να επιχειρηματολογήσουμε όταν θα βρεθούμε ε, καθήμενοι απέναντι στο, από το Συμβούλιο και θα πρέπει τα επιχειρήματα να τα προβάλλουμε και στον Ευρωπαίο πολίτη γιατί το μόνο που μπορεί να επηρεάσει ε, τους και τους ηγέτε. είναι είναι η κοινή γνώμη. Άρα να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να γίνουμε κατανοητοί από τους συμπολίτε μας, από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ήταν μια εξαιρετικά καλή συζήτηση. Ευχαριστώ τους εισηγητές, τους συνεισηγητές, τους εκπροσώπους εισηγητές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση στις 2.30 θα ξαναβρεθούμε για συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών, η οποία ενδεχομένως να μας επιτρέψει να άρουμε μία επιφύλαξη που είχαμε καταθέσει κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ε, οφείλω να διευκρινίσω το εξής. Σε ό,τι αφορά στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τροπολογίε για την ενδιάμεση έκθεση πρέπει να κατατεθούν το αργότερο στις 6 ώρα το απόγευμα στις 15 Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή των Προπολογισμών θα λάβει χώρα στις 5 Νοεμβρίου και στην πρώτη Ολομέλεια του Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει στο Στρασβούργο και θα αποφανθεί. Ε, τη λήξη της πρωινής μας συνεδρίασης.